Liebe Kolleginnen und Kollegen. Συνάδελφοι, ας ξεκινήσουμε γιατί έχουμε καθυστερήσει ήδη 10 λεπτά. Θεωρήσαμε ότι η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Απασχόλησης ε, θα είχε φτάσει. Θα έρθει σίγουρα, αλλά ας ξεκινήσουμε εμείς γιατί αλλιώς ε, θα μας τελειώσει ο χρόνος. Λοιπόν, σας καλωσορίζω όλους στην σημερινή μας ακρόαση την οποία και διοργανώνουμε από κοινού με την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Σήμερα επιλέξαμε ένα ιδιαίτερα περίπλοκο θέμα, το οποίο έχει προκαλήσει και διαφωνίες και το οποίο βεβαίως έχουμε συζητήσει αρκετές φορές εδώ στην Επιτροπή μας. Α, ήρθε. Σε καλωσορίζω, Μαϊτα Ουλσκουκ θα μας παρουσιάσει σήμερα στην Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας ε, την έκθεσή της για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης η Helga Truppel, μετά την ακρόαση όμως. Επίσης θέλω να καλωσορίσω θερμά τον Επίτροπο Τίμπορ Ναύρατσιτς, του οποίου η παρουσία θεωρώ ότι τονίζει την ιδιαίτερη σημασία που έχει για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Επίσης θα έχουμε την ευκαιρία στο πλαίσιο της ακρόασης να παρακολουθήσουμε και μια παρουσίαση μιας μελέτης που εκπώνησε το Τμήμα Πολιτικής Β για αυτό το θέμα. Τα συμπεράσματα αυτής της δημόσιας ακρόασης πιστεύω ότι θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμα και θα βοηθήσουν και την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας και την Επιτροπή Απασχόλησης. Έχουμε μια σειρά από εξαίρετους εμπειρογνώμονες ε, ως προσκεκλημένους εδώ ε, οι οποίοι καλύπτουν διάφορους τομείς της κοινωνίας των πολιτών αλλά και διάφορες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που εργάζονται στον τομέα του εθελοντισμού. Έχουμε μαζί μας λοιπόν τον κύριο Ζήμον Μπροκ από το Ockham Institute for Policy Support που θα μας ε, παρουσιάσει την μελέτη της, ε, του Τμήματος Πολιτικής. Επίσης, να καλωσορίσω τον κύριο Μάνφρετ Φον Χέμπελ από την Γερμανική Εθνική Υπηρεσία για το πρόγραμμα Erasmus Plus που θα μας παρουσιάσει την, προοπτική, την οπτική των εθνικών υπηρεσιών. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Πάβελ Τράντινα, που είναι πρόεδρος του Τμήματος Απασχόλησης Κοινωνικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Έχουμε μαζί μας την κυρία Γκαμπριέλα Σίβικο που είναι Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Εθελοντισμού, τον κύριο Πιότρε Σαντόφσκι που είναι Γενικός Γραμματέας του Volont Europe που θα μας ε, παρουσιάσει ορισμένες ευκαιρίες και προκλήσεις για την κινητικότητα των νέων, το Erasmus και το, την εθελοντική εργασία όσον αφορά τον, ε, το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Κώστα Μοσχοχωρίτη, ελπίζω να το είπα καλά, κάπως καλά, που είναι Γενικός Γραμματέας του Ίντερ ε, ΣΟΣ, που θα φωτίσει το ζήτημα των προκλήσεων όσον αφορά τον εθελοντισμό και τον επαγγελματισμό και τέλος έχουμε μαζί μας την κυρία Άννα Βίντεγκρεν, Γενική Γραμματέα του Ευρωπαϊκού ε, Φόρουμ Νεότητας, που θα ε, μας ε, μιλήσει για το ποια θα είναι τα ωφέλη αυτού του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης για την, για την νεολαία στην Ευρώπη. Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε γεμάτο πρόγραμμα σήμερα το απόγευμα. Να σας καλωσορίσω όλους άλλη μια φορά. Για να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο για τη συζήτηση. Θα ήθελα να καλέσω όλους τους προσκεκλημένους να τηρήσουν το χρόνο ομιλίας που θα τους ε, ε, Έχετε ο καθένας σας πέντε λεπτά. Σας είχαμε άλλωστε αποστείλει και ένα ερωτηματολόγιο το οποίο ε, απαντήσατε όλοι με πολλές πληροφορίες και τις απαντήσεις σας άλλωστε τις έχουμε διαβιβάσει και σε όλα τα μέλη της Επιτροπής και μπορεί η συζήτηση να περιστραφεί και γύρω από τις απαντήσεις αυτές. Πρωτού ξεκινήσουμε με τις παρουσιάσεις, θα ήθελα να δώσω την, ε, το λόγο και στην κυρία Ουλσκοκ, που είναι πρόεδρος της Επιτροπής Απασχόλησης, στον ε, Επίτροπο Ναύρατσιτς, αλλά και την συγγήτρια της Επιτροπής Πολιτισμού, την Χέλγα Τρούπελ, Πρώτον, ε, ας ξεκινήσουμε με την ε, κυρία Ουλφσκοκ. Ευχαριστώ Πέτρα και εγώ καλωσορίζω όλους συμμετέχοντες, κυρίως τους ε, εμπειρογνώμονες που θα συνεισφέρουν με πολύτιμο τρόπο στην ακρόαση για όλους μας εκφράζοντας απόψεις περιστόχων και αποτελεσματικότητας του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης ανήκει σε μια πρωτοβουλία που θα δίνει ευκαιρίες στους ε, νέους να συμμετέχουν σε δραστηριότητες αλληλεγγύης, συμπεριλαμβανομένης μαθητείας, εργασίας και προφανώς αυτό είναι κάτι που θα έχει θετικές ε, συνέπειες διότι θα βελτιώσει την απασχολησιμότητα και θα διευκολύνει την μετάβαση προς την κανονική απασχόληση. Αυτό που θα ήθελα υπογραμμίσω σήμερα είναι ότι 35 εκατομμύρια ευρώ από τον προϋπολογισμό διατίθενται για τη χρηματοδότηση αυτού του σώματος από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Και η πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ε, μετακίνηση των πόρων από τα προγράμματα ε, καινοτομίας, περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία χρειάζονται ούτως ώστε να εξυπηρετήσουν τους υφιστάμενους σκοπούς και δεν θα πρέπει να δεχθούν πιέσεις. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν τα χρήματα με τον αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο και αποτελεσματικότητα σημαίνει θέσεις απασχόλησης και μέλλον για τους νέους της Ευρώπης που δεν έχουν κάποια θέση. Τώρα προσπαθούν να βρουν μια δουλειά, προσπαθούν να βρουν μια θέση στη ζωή τους όπου να είναι ικανοποιημένοι και να αισθάνονται ότι υπάρχει ένα νόημα στη ζωή τους, ότι είναι χρήσιμοι. Ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Με ενδιαφέρον θα ήθελα να ακούσω τι έχουν να, πει, να πούν οι εμπειρογνώμονες και όλοι όσοι ήρθατε για να συμμετάσχετε σε αυτή την συνεδρίαση. Καλώς. Λοιπόν, εσείς έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ Μαρίτα για τα εισαγωγικά σου λόγια αυτά. Χωρίς περαιτέρω χρονοτριβή θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Επίτροπο Ναύρατσιτς. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο για περίπου 10 λεπτά, όχι παραπάνω. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι. Σε πρόσφατη ομιλία του για την κατάσταση στην Ένωση, ο Πρόεδρος κύριος Γιούνκερ είπε ότι ήταν ιδιαίτερα υπερήφανος για τους νέους που υπηρετούν στο νέο αυτό σώμα αλληλεγγύη, στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύη, Δίνουν αλληλεγγύη στη ζωή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτά είπε. Εξίσου είμαι περήφανο διότι από όταν ξεκίνησε αυτή η δραστηριότητα το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύη πέρσι, πάνω από 38.500 νέοι άνθρωποι έχουν δηλώσει εθελοντέ. Όλοι από αυτοί είναι έτοιμοι να προσφέρουν συντροφιά στους ε, μοναχικούς ανθρώπους, ε, να βοηθήσουν τους πρόσφυγες που έχονται στην Ευρώπη, να καθαρίσουν ε, μολυσμένες ακτές ή να βοηθήσουν κοινότητες με άλλους τρόπους. Είναι το πρώτο βήμα προς τη φιλοδοξία μας που έχουμε το ώστε στο 2020 να έχουμε 100.000 νέους Ευρωπαίους που θα έχουν τη δυνατότητα να βοηθήσουν εκεί που υπάρχει ανάγκη βοηθείας περισσότερο. Το 2017 περιμένουμε να δώσουμε πάνω από 16.000 θέσεις για εθελοντική εργασία και 3.600 ε, νέοι θα μπορέσουν να δραστηριοποιηθούν επί τόπου πριν το τέλος του έτους. Περίπου 1.800 ήδη ξεκίνησαν την τοποθέτησή τους και οι αριθμοί αυτοί αυξάνονται. Τον περασμένο μήνα ο πρόεδρος Αντώνιο Ταγιάννη και εγώ επισκέφθηκα τους εθελοντές στην Νόρτσα, στην Ιταλία, σε μια πόλη, σε μια περιοχή που προσπαθεί να ανακάμψει από πολλούς καταστροφικούς σεισμούς που συνέβησαν πέρσι. Εκεί είδαμε ότι είναι αποφασισμένοι αυτοί οι νέοι που συμμετέχουν σε αυτό το σώμα αλληλεγγύης να βοηθήσουν τους κατοίκους να ανοικοδομήσουν τις κατοικίες τους και να ξαναβρούν τη ζωή τους. Αυτό είναι ένα συγκινητικό σημάδι ελπίδας. Σας καλώ να συμμετάσχετε στις διαπραγματεύσεις για το προτινόμενο κανονισμό για το σώμα αλληλεγγύης στο ευρωπαϊκό, στο ίδιο πνεύμα, με την ίδια δέσμευση ε, που δείχνουν, ε, αφοσίωση που δείχνουν για αυτοί οι νέοι που έχουν μπει σε αυτό το σώμα. Συζητήσεις με τους νέους και τους εμπλεκομένους φορείς τον τελευταίο μήνα, τελευταίους μήνες, είδα ότι υπάρχουν πολλές δυνατότητες να κινηθούμε προ το μέλλον γρήγορα. Τώρα, πώ προτιθέμεθα να πετύχουμε του στόχου μα για το Ευρωπαϊκό Αυτό Σώμα το σχέδιο του κανονισμού συγκεράζει όλε τι δραστηριότητε που είναι κατακαιρματισμένε μέσω οκτώ προγραμμάτων. Αυτή η προσέγγιση έχει αρκετά ωφέλη. Καταρχά θα παράσχουμε σαφείς συνεκτικούς κοινού λόγους, συνθήκες και όρους, μαζί με μια πύλη που θα είναι ένα σημείο εισόδου με εύκολη πρόσβαση στον θελοντισμό, στην μαθητεία και στις ε, ευκαιρίες για απασχόληση. Ε, δεύτερον, αυτό σημαίνει περισσότερη χρηματοδότηση και περισσότερες μορφές εθελοντισμού για να επιλέξει κανείς. Και τρίτο, θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε να συμμετάσχουν εκείνοι που δεν μπορούν να καλυφθούν τα τρέχοντα προγράμματα. Αυτό δείχνει σαφέστατα λοιπόν ότι η προσέγγιση μας είναι πραγματικά επικεντρωμένη στις ανάγκες των νέων. Θα διερωτάστε γιατί δεν έχουμε καθορίσει όλα τα στοιχεία στον κανονισμό με, με αυστηρότητα και περιορισμένα. Έχουμε κάθε λόγο. Θα μας συμμετέχοντε κάθε δυνατότητα επιλογής να υποστηρίξουν διάφορες κοινότητες και να συμβάλλουν και τον τρόπο στην κοινωνική συνοχή στην Ένωσή μας. Γι' αυτό το λόγο έχουμε και την αλληλεγγύη, δραστηριότητα αλληλεγγύη. Προσπαθούμε να ορίσουμε αυτή την έννοια. Η δραστηριότητα αλληλεγγύη, το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύη μπορεί πραγματικά να απογειωθεί και να κινηθεί αν έχουμε ευρύ φάσμα νέων που συμμετέχει και διαφόρων οργανώσεων. Κανεί δεν πρέπει να αποκλείεται εξ αρχή, διότι ο κανονισμό καθορίζει διάφορου ορισμού που θα είναι περιοριστικοί οι ε, οργανώσεις των κατοίκων του πληθυσμού θα πρέπει να δουν πώς θα καλύψουν τις ανάγκες τους και να βρουν τον καλύτερο τρόπο να βρουν τη θέση τους στο μελλοντικό σχήμα που θα έχει αυτό το σώμα αλληλεγγύης. Αλλά είστε βέβαιοι ότι μέσω αυστηρών ποιοτικών ελέγχων θα εξασφαλίσουμε ότι όλες οι δραστηριότητες είτε προτείνονται από τους νέους είτε από οργανώσεις και φορείς θα εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Πιο συγκεκριμένα θα εξασφαλίσουμε ότι δεν θα οδηγήσουν σε αντικατάσταση θέσεων εργασίας. Οι εθελοντικέ δραστηριότητε που οργανώνονται στα πλαίσια του Σώματο Αλληλεγγύη θα εδράζονται επί της πλούσιας εμπειρία που έχουμε οικοδομήσει ε, με την, την υπηρεσία εθελοντισμού την ευρωπαϊκή και ε, τα προγράμματα μαθητείας θα εντάσσονται στην κατάρτιση και θα πρέπει τις απασχόλησεις να ταιριάζουν με τους εθνικούς κανόνες περί εργασίας. Όλα αυτά έχοντας τα υπόψη. Απευθυνόμεθα προ όλου του νέου και με εκείνου που έχουν λιγότερε ευκαιρίε. Αυτό πιστεύω ότι είναι μία από τι προτεραιότητέ μου και γι' αυτό έχουμε σχεδιάσει ένα φάσμα νέων ε, μορφών εθελοντισμού θέλω να προσφέρουμε. Βραχυπρόθεσμε δραστηριότητε που διαρκούν μεταξύ δύο εβδομάδων και δύο μηνών ε, θελοντικές ομάδες που θα παρέχουν καλύτερο περιβάλλον για ομάδες, ε, τοποθετήσεις μέσα στη χώρα ε, και διάφορα προγράμματα ελεγγύη. Θα διαθέσουμε και άλλους πόρους να πληρώνουμε για συνοδεία ανθρώπων ή για το κόστος διαφόρων μέσων που χρειάζονται άτομα με αναπηρία. Γνωρίζω πλήρως ότι οι διάφορες οργανώσεις εθελοντών έχουν πολύ σημαντικό ρόλο για να βοηθήσουν επίσης και νέους με προβλήματα. Ε, θα συνεχίσουν να παίζουν το ρόλο του στα πλαίσια του σώματος αλληλεγγύης. Το σώμα θα δίνει στους νέους συμπληρωματική πρόσβαση σε φορείς που έχουν ετικέτα ποιοτική και που είναι καταγραμμένοι και καταχωρημένοι οι φορείς αυτοί στην ε, πύλη. Αυτή η νέα θηρίδα θα πλουστεύσει τη συμμετοχή. Κατά πολύ. Τόσο αφορά τον προπολογισμό, θέλω να είμαι σαφέστατος, Πιστεύω πως και εσείς ότι οι νέες ιδέες χρειάζονται και φρέσκο χρήμα. Και γι' αυτό η πρότασή μας προϋπολογισμού περιλαμβάνει 86,5 εκατομμύρια ευρώ νέων πόρων. Αυτό αντιπροσωπεύει 25% του συνολικού προϋπολογισμού που είναι 341,5 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά τα νέα χρήματα, 70 εκατομμύρια ευρώ θα δώσουν τη δυνατότητα ουσιαστικά να αυξήσουμε τον αριθμό των ευκαιριών για εθελοντισμό για την περίοδο από το 2018 μέχρι το 2020. Από τα αρχικά που είχαμε προβλέψει 40.000 το Erasmus Plus στα, 77.800 εντός του πλαισίου του σώματος και του Erasmus Plus. Λοιπόν, το Σώμα Αλληλεγγύης δεν θα υπονομεύσει άλλες πρωτοβουλίες νεότητας που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Νεολαίας του Erasmus Plus. Αντιθέτως, ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μια συμπλήρωση πόρων στο Erasmus Plus στα πλαίσια της ενδιάμεσης αναθεώρησης του τρέχοντος πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας για την σταθερή υποστήριξή σας, ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε ότι ο Erasmus Plus θα έχει τους αναγκαίους πόρους που χρειάζεται και αξίζει. Ευχαριστώ την Επιτροπή Πολιτισμού ε, που, πρότεινε, που υποστήριξε την αύξηση την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2018 και που ζήτησε συμπληρωματικού ε, πόρου. Ε, όσον αφορά το Σώμα Αλληλεγγύης, το σχέδιο του κανονισμού προτείνει να διατεθούν το 80% των πόρων σε εθελοντικές δραστηριότητε και 20% σε μαθητείες και θέσεις εργασίας. Αυτή η ενδεικτική κατανομή θα μας δώσει την ευελιξία να προσαρμοστούμε στις ανάγκες και τα συμφέροντα των νέων και των οργανώσεων κατά τη διάρκεια ζωής του προγράμματος. Ε, μια άλλη πτυχή που είναι σημαντική για μένα είναι η συνεργασία με παρόμοια σχήματα και προγράμματα εντός των ε, κρατών μελών, όπως ε, η υπηρεσία σε πολιτικό επίπεδο, η στήριξη πολιτών και θα δώσουμε ε, πρόσβαση στα εθνικά σχήματα στην πύλη αυτή και θα παράσχουμε υποστήριξη όπως είναι η μαθητεία, η ασφάλιση και η κατάρτιση. Κυρίε και κύριοι, το να βοηθάμε τους άλλους είναι σαν να ρίχνουμε ε, μια πέτα στο νερό, δημιουργούνται κυματάκια στο νερό και οι εθελοντές στην Όρτσα και χιλιάδες άλλοι που θα δραστηριοποιηθούν σε όλη την Ευρώπη δίνουν πνοή ζωής σε διάφορες κοινότητες, δημιουργούν νέες φιλίες και βοηθούν να οικοδομηθεί μια κοινωνία που είναι πιο συνεκτική και ενώ βοηθούν τους άλλους επίσης κερδίζουν ε, και νέες δεξιότητες και βλέπουν τα πράγματα με άλλα μάτια και μπορούν να απτυχθούν και να εκμεταλλευτούν στο μέλλον καλύτερα τα ταλέντα τους στην μελλοντική τους προσωπική και επαγγελματική ζωή. Έχω την πεποίθηση το σχέδιου κανονισμού δημιουργεί τις ηθίκες εκείνες για μια κοινότητα ανθρώπων που έχουν παρόμοια νοοτροπία να συνδεθούν και να προχωρήσουν μαζί μπροστά. Σημαίνεται πρέπει να τους δώσουμε όμως το χώρο να στερνιστούν τις αρχές του σώματος αλληλεγγύης, να ρίξουν ιδέες, να μοιραστούν εμπειρίες να δημιουργήσουν προγράμματα μαζί και να εμπνεύσουν και νέους και νέα μέλη. Το Σώμα Αλληλεγγύης θα επιτρέψει τους νέους από όλη την Ευρώπη να συμμετάσχουν στην οικοδόμηση κοινοτήτων μέσω πλατφορμών ε, online, κοινωνικών ε, ε, μέσων δικτύωσης και μέσω του κανονισμού μπορούμε να φτιάξουμε τα θεμέλια για, μια, για ένα πραγματικό ευρωπαϊκό κίνημα αλληλεγγύης. Κλείνοντας ευχαριστώ του συζητητές και όλα τα μέλη που συμμετέχουν στην νομοθετική διαδικασία. Ευχαριστώ για τι προσπάθειε που κάνετε και την αφοσίωση που δείχνετε για την νέα πρωτοβουλία. Η επίτευξη, μια ταχεία επίτευξη πολιτική συμφωνία θα είναι υποφελή για πολλού νέου στην Ευρώπη που είναι πρόθυμοι να κάνουν τη διαφορά και προσβλέπω στο να ακούσω τι απόψει σα. κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην ε, Χέλγα Τρούπελ που είναι η συγγήτρια της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας. Χέλγα, πολύ σύντομα, ευχαριστώ πολύ Πέτρα. Είναι σαφές ότι έχουμε σήμερα την ακρόαση, αλλά εγώ έχω υποβάλει την έκθεσή μου από τις 19 Σεπτεμβρίου. Αυτό σημαίνει ότι είμαι ανοιχτή στο να ακούσω βεβαίω όλου του συναδέλφου και του εμπειρογνώμονε και βεβαίω θα είμαι έτοιμη να τροποποιήσω και την έκθεσή μου, αν πιστώ ε, ότι υπάρχει τέτοια ανάγκη. Το λέω αυτό ε, για να σας πω ότι ε, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική η ακρόαση που διοργανώνεται σήμερα. Απλώς λόγω χρονοδιαγράμματος ε, ήμουν αναγκασμένη να υποβάλω την έκθεσή μου ήδη από τις 19 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα όλη η ομάδα μου και το επιτελείο μου εργάστηκε όλο το καλοκαίρι πολύ σκληρά για να επιτύχουμε αυτό το στόχο. Τώρα, δεν θέλω να ε, υπησέλθω σε πολλές λεπτομέρειες, απλά θέλω να τοποθετηθώ πολιτικά εντάχει γύρω από ε, το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Νομίζω ότι η πρόταση του Juncker για τη δημιουργία αυτού του σώματος είναι πολύ καλή ιδέα. Και είναι προφανές ότι ο πρόεδρος προσπαθεί να βρει άλλο ένα εμβληματικό πρόγραμμα όπως το Εράσμους ε, διότι φαίνεται ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει έλλειψη αλληλεγγύης σε πολλά επίπεδα. Την ενστερνίζομαι λοιπόν την ιδέα αυτή θεωρώντας όμως ότι πρέπει να τη βελτιώσουμε. Δεν θέλω να την κατεπολεμήσουμε, απλά θέλω να τη βελτιώσουμε. Υπάρχουν τρία πράγματα που θέλω να βελτιώσουμε. Πρώτον, το όνομα. Νομίζω το, όρο όρος σώμα, κορ, και στα γερμανικά αλλά και σε πολλές γλώσσες ε, δεν ηχεί ε, ιδιαίτερα όμορφα. Ε, γι' αυτό θα ήθελα να, ε, αντί για σώμα να χρησιμοποιούμε τον όρο πρωτοβουλία. Δεύτερον, για τον προπολογισμό. Ο Επίτροπο έχει δίκιο. Υπάρχουν 80 εκατομμύρια ε, αδιάθετα κονδύλια. Εσείς τα είπατε φρέσκο χρήμα. Δεν είναι ακριβώς φρέσκο χρήμα. Είναι χρήματα τα οποία δεν έχουν διατεθεί ε, στα κράτη-μέλη. Αν πράγματι όμως θέλετε ε, να απογειωθεί όπως είπατε αυτό το νέο πρόγραμμα χρειάζεται πραγματικό φρέσκο ε, χρήμα. Και γι' αυτό σας καλώ να καταβάλλετε προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση. Δεύτερον, τρίτον μάλλον, πιστεύω ότι πραγματικά πρέπει το πρόγραμμα αυτό να ωφελήσει νέους ανθρώπους που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση. Γιατί εμείς εδώ ερχόμαστε πολύ συχνά σε επαφή ε, με ασκούμενους οι οποίοι είναι κοσμοπολίτες, έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση κτλ. Είμαστε λίγο σε μια φούσκα εδώ μέσα. Ε, υπάρχουν όμω εκατομμύρια νέοι άνθρωποι οι οποίοι καθόλου δεν έχουν αυτέ τι ευκαιρίε όπω οι νέοι που βρίσκονται εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και νομίζω ότι πρέπει να, τεθεί, να τεθεί και αυτή, αυτή η πληθυσμιακή ομάδα στο επίκεντρο. Και τελευταίο, αναφερθήκατε στην, ε, στην απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων. Γνωρίζουμε όλοι ότι η νεανική ανεργία είναι υπερβολικά υψηλή σε πάρα πολλά κράτη-μέλη και πρέπει να καταπολεμηθεί. Όμως, αν προχωρήσουμε όπως προτείνεται, δηλαδή χωρίς να υπάρχει ε, διάκριση μεταξύ του εθελοντισμού και των δραστηριοτήτων αλληλεγγύης αφενός και αφετέρου από την, τις δραστηριότητες απόκτησης επαγγελματικών δεξιοτήτων μπορεί το μείγμα αυτό να είναι εκρηκτικό. Αν υπάρχει σαφής ορισμός ώστε να ε, αποφύγουμε κάθε κατάχρηση από την αγορά εργασίας και να αποφύγουμε κάθε περίπτωση κατά την οποία ενδέχεται νέοι άνθρωποι να πληρώνονται λιγότερα χρήματα από ό,τι θα έπρεπε κανονικά να λαμβάνουν υπό την πρόφαση ότι ασκούν εθελοντισμό, τότε αν αποφύγουμε λοιπόν αυτό, τον κίνδυνο, ε, νομίζω ότι τότε μόνο θα επιτύχουμε τους πραγματικούς στόχους. Αλλιώς καλύτερα να απαλλαγούμε πλήρως από αυτήν την επαγγελματική διάσταση του σώματος αλληλεγγύης. Ευχαριστώ πολύ και με αυτό περνάμε στην ε, συζήτηση. Θα δώσω το λόγο στον ε, εισηγητή της Επιτροπής Απασχόλησης, τον κύριο Μπόνιφαϊ, για δύο με τρία λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, ξεχάσατε ότι είμαι και εγώ ο μιλητής στο πάνελ, είμαι και εγώ εισηγητής, ξέρετε. Άλλωστε ε, γνωρίζετε ότι τα ζητήματα της απασχόλησης είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας Επιτροπής Απασχόλησης. Χαίρομαι λοιπόν που βρίσκομαι εδώ, γιατί νομίζω ότι και αυτά τα θέματα που έθεσε η συνάδελφος, που τα έχουμε ξανασυζητήσει και στο παρελθόν, είναι ακριβώς το σημαντικότερο θέμα. Πρέπει να το δούμε σε λεπτομέρειες και να δούμε αν μπορούμε να βρούμε λύση σε αυτό το θέμα. Και θέλω εισαγωγικά να προσθέσω κάτι. Καταρχάς να ευχαριστήσω ε, όλους τους ε, προσκεκλημένους, τον Επίτροπο που παρίσταται εδώ, την, τις Προέδρους ε, κυρία Κάμερβερτ και Ουλφσκοκ που εκπροσωπεί τον, τον πρόεδρο της δική μα επιτροπή για αυτή τη συζήτηση που γίνεται σήμερα. Ο χρόνος μα είναι περιορισμένος πράγματι, αλλά ε, έχουμε πολλά σημαντικά θέματα να συζητήσουμε. Όπως είπε και η συνάδελφος, υπάρχει το θέμα των χρημάτων, της χρηματοδότησης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Συμφωνώ ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε αν μπορούμε να ε, δεσμεύσουμε περισσότερα χρήματα από τα κράτη-μέλη με πραγματικό φρέσκο χρήμα δηλαδή για το πρόγραμμα αυτό αφενός και βεβαίω είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι έχουν υπάρξει ήδη 37.000 εγγραφές στην online πύλη. Ε, είναι πράγματι πολύ ενθαρρυντικό σημαντικό αυτό το στοιχείο, ε, ιδίως έχοντας κατά νου το στόχο περί 100.000 εγγραφών έω το 2020, όπως τον προσδιορίσε ο πρόεδρος Γιούγκερ. Ωστόσο, ε, πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτόν τον κίνδυνο της υποκατάστασης πραγματικών θέσεων εργασία με εθελοντική δουλειά. Άρα πρέπει να οριοθετήσουμε σαφώς... Ε, τι ακριβώς και με ποιον ακριβώς τρόπο μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση σε αυτό το σώμα αλληλεγγύης και εθελοντισμού και στο πλαίσιο αυτό έχουμε ήδη συζητήσει με τη συνάδελφο Τρούπελ ε, τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα χρήματα που έχουν προέλθει ε, μάλιστα και από άλλα προγράμματα. Εγώ προσωπικά είμαι πεπισμένος ότι μπορούμε να βρούμε συμβιβασμό ώστε να διατηρηθεί και αυτή η επαγγελματική διάσταση με έναν τρόπο ε, που θα εξασφαλίζει ε, ότι θα υπάρχει και θα αξιοποιείται όλη η εμπειρογνωμοσύνη την οποία θα ακούσουμε και σήμερα εδώ. Διότι νομίζω ότι ε, κάνουμε κάτι λίγο διαφορετικό σε σχέση με το παρελθόν. Άρα χρειάζεται μια προστιθέμενη αξία. Αφενός χρειάζεται άμεση πρόσβαση, ακόμη και αν είμαστε όλοι πολύ ενωμένοι ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, λέγοντας ότι χρειάζεται να διατηρήσουμε την εμπειρογνωμοσύνη ε, και τις γνώσεις όλων των ενδιάμεσων οργανώσεων, πρέπει να ξεκαθαριστεί σαφώς αυτό και στο επίπεδο της συμμετοχής στο πρόγραμμα αυτό. Και τέλος, σχετικά με το θέμα του ποιε οργανώσεις θα επιτρέπεται να συμμετέχουν ε, προσφέροντας και ευκαιρίες απασχόλησης. Η σύνδεση του εθελοντισμού με την απόκτηση εμπειρίας είναι δυνατή, είναι εφικτή, χωρίς απαραίτητα όμως να, να καταλήγουμε σε καταστάσεις που ενδεχομένως να ε, ε, υπόκεινται σε πολύ αυστηρή κρατική από όσου μας παρακολουθούν. Ε, και νομίζω ότι για να το κάνουμε αυτό χρειάζεται μια πολύ συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, όλων των επιτροπών, όλων των συναδέλφων. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Και τώρα θα ακούσουμε την παρουσίαση της μελέτης που εκπώνησε το Τμήμα Πολιτικής, Ευρωπαϊκό Σώμα και Εθελοντισμός, είναι ο τίτλος αυτής της μελέτης. Να καλωσορίσω άλλη μια φορά τον κύριο Ζήμον Μπρουκ που θα μας παρουσιάσει την μελέτη αυτή. Το να παρουσιάσω τα βασικά πορίσματα στην δελεχούς αναλύσεως της νομοθετικής προτάσεως για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Αυτή η ανάλυση διεξήχθη από τον υποφαινόμενο και συνάδελφο κύριο Πάσκου ε, για την Επιτροπή Πολιτισμού της, ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στεστήκαμε επί τριών πτυχών που είναι οι βασικοί τομείς Πρώτα απ' όλα, με ποια έννοια θα προσθέσει αξία αυτό το σώμα θελοντών σε επίπεδο κοινωνία, ποιε είναι οι προκλήσει όταν αφορά να συνδεθεί με το Erasmus Plus και άλλα προγράμματα τη Ευρωπαϊκή Ενώσης και πώ μπορεί αυτό το Ευρωπαϊκό Θελοντικό Σώμα να λειτουργήσει με έναν τρόπο που συμπληρώνει και δεν αντικαθιστά την επιπληρωμή εργασία, την αμοιβόμενη εργασία. Λοιπόν, για να απαντήσω αυτή τη ερωτήσεις, η μελέτη εδράζεται επί έρευνας ε, θεωρητικής και επί συνεντεύξεων. Ε, Καταρχά εν συντομία, να κάνουμε εισαγωγή ποιο είναι ο, βασικό στόχο και σε ποια υπόθεση βασιστήκαμε. πώ θα οδηγήσει σε αποτελέσματα ο Ευρωπαϊκό Σώμα όπω Όπως γνωρίζετε, ο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύη γενικό στόχο έχει να αυξήσει τη συμμετοχή των νέων και οργανώσεων νέων με ένα προσβάσιμο και σε προσβάσι... με προσβάσιμο τρόπο σε ποιοτικέ δραστηριότητε αλληλεγγύη, να ενισχυθεί η συνοχή και η αλληλεγγύη στην Ευρώπη, να υποστηριχθούν κοινότητε και να ανταποκριθούν σε προβλήματα τη κοινωνία. Έτσι, οι νέοι ηλικία 18 μέχρι 30 ε, μπορούν να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες αλληλεγγύης διασυνοριακά και εντός χωρών όπως τοποθετήσεις επιτόπου, ομάδες, διάφορα προγράμματα, δικτύωση και επίσης θα δίνεται και ποιοτική, ε, ε, ποιοτικό σήμα σε διάφορους οργανισμούς. Λοιπόν, μέσω συγκέντρωση θεωρητικών δυνατοτήτων από προγράμματα που υπάρχουν τώρα και συλλογικά οι θεωρητικέ δραστηριότητε να έχουν ένα κοινό τίτλο, η ζήτηση και η προσφορά μπορεί να ταιριάξουν καλύτερα. Ο συντονισμό δίνει αποτελέσματα. Δηλαδή, περισσότεροι νέοι θα συμμετάσχουν σε δραστηριότητε αλληλεγγύη και θα παρέχουν ποιοτικέ υπηρεσίε και τα αποτελέσματα συνεπώ θα είναι καλύτερα στις διαβουλεύσεις είδαμε ότι υπάρχει μια γενική εκτίμηση για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Σώματος ε, θελοντισμού από τους εμπλεκόμενους φορείς και είδαμε ότι υπάρχουν και θετικά στοιχεία από τη μελέτη που κάναμε στην πρόταση. Δηλαδή αυτό το σώμα μειώνει τους φραγμούς που έχουν εντοπιστεί για τα άτομα να κάνουν δραστηριότητες εθελοντισμού, κυρίως η παροχή ε, πληροφοριών, υποστήριξη για ανθρώπους, για νέους που έχουν προβλήματα συμπεριλαμβάνοντα επίση τη μαθητεία, τα στάζ και τις θέσει απασχόληση και τις διάφορε άλλε δράσει αλληλεγγύη και διευρύνεται έτσι το πεδίο εφαρμογή και δραστηριοποίηση του εθελοντισμού στην Ευρώπη. Δεύτερον, η εισαγωγή της ε, ετικέτα ποιότητα μπορεί να δημιουργήσει μια οτροπία ποιοτική, αν δεν υπάρχει ήδη. Και αυτό το σώμα, συγκρίσει με άλλε μορφέ εθελοντισμού, μπορεί να παράσχει ίσε ευκαιρίε ε, για όλου του νέου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανεξάρτητα από τι ε, δυνατότητε που δημιουργούνται σε εθνικό επίπεδο. Παρά τα θετικά στοιχεία εντοπίσαμε όμω και κάποιε ανησυχίε και προβλήματα. Μπορούν να μοδοποιηθούν σε πέντε κατηγορίε που θα συζητήσω ξεχωριστά και θα παράσχω και κάποιε συστάσει. Λοιπόν, αν δείτε πρώτα απ' όλα, σχετίζεται με την αρχή των ε, συμπράξεων. Δηλαδή, όταν οι μπλεκόμενοι φορείς ε, συμμετέχουν επαρκώς ε, με ποιοτικό τρόπο σε αυτό το σώμα και να προωθούν τα συμφέροντα, κατά πώς τα συμφέροντα και των οργανώσεων, των κοινωνικών εταίρων και των εθελοντών εκπροσωπούνται όταν δημιουργείται το πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Εθελοντισμού και συστήνεται να δοθούν και συγκεκριμένε κατευθύνσει στην πρόταση σχετικά με τη συμμετοχή των μπλεκομένων φορείων στο σχεδιασμό, παρακολούθηση και υλοποίηση των στόχων, για να δούμε και ποια είναι τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται. Οπότε είναι πολύ χρήσιμο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη-μέλη, οι εθνικοί οργανισμοί να συνεργάζονται στενά και σε σύμπραξη με τα συνδικάτα και με κυβερνητικέ οργανώσει, με οργανώσει νέων και άλλου φορεί που είναι υπεύθυνοι για την πρόθεση των δραστηριοτήτων αλληλεγγύη. Τώρα σχετικά με, τον, με τους στόχους εντοπίσαμε τρεις ανησυχίες. Κατά πόσο αυτό, το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης μπορεί να πετύχει τις 100.000 αυτές τις δραστηριότητες αλληλεγγύης την τριετία. Όλοι γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εθελοντισμού ε, έχει, πέρασε 20 χρόνια να φτάσει σε αυτό το επίπεδο και η παρούσα πρόταση δεν εξηγεί επακριβώ πώ το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύη θα μπορέσει να φτάσει σε αυτό το στόχο και πώ θα μπορέσει να βρει επαρκή επαρκή, επαρκή ποιοτική συμμετοχή. Υπάρχει και άλλη ανησυχία κατά πόσο όλες οι φυστάμενες και νέες δράσεις θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη συμμετοχή όσον αφορά των ε, ομάδων που έχουν προβλήματα. Διότι ε, το, ε, ήδη οι οργανώσεις θα μπορέσουν, θα, θα συμμετάσχουν, κατά πόσο θα βρούνε και τη δυνατότητα νέοι με προβλήματα να συμμετάσχουν. Λοιπόν, τελευταία ανησυχία όσον αφορά αυτό το θέμα είναι κατά πόσο το Ευρωπαϊκό Σώμα αυτή η δημιουργεί διαφορέ μεταξύ διαφόρων εθελοντών που κάνουν την ίδια δουλειά σε διαφορετικά προγράμματα. Οι εθελοντέ οι οποίοι δεν χρηματοδοτούνται από αυτό το σώμα αλλά θα εργάζονται εντό του ίδιου οργανισμού δεν θα έχουν πιστοποιητικό μέσω του οποίου θα φαίνεται ότι έχουν αποκτήσει δεξιότητε και ίσω το δικό του πιστοποιητικό να μην έχει την ίδια αξία. Σα σύσταση λοιπόν, το, η πρόταση για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύη θα πρέπει να διευκρινίσει πώς λειτουργεί συμπληρωματικά με εθνικές πρωτοβουλίες και πώς οι εθνικές πρωτοβουλίες μπορούν να ωφεληθούν από τον Ευρωπαϊκό Φορέα, κυρίως μέσω της θέσπισης δράσεων εντός μιας χώρας, δράσεων αλληλεγγύης. Πρέπει να επαναξεταστεί πώς οι εθελοντές που δεν ανήκουν στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης μπορούν να εξυπηρετηθούν από το μηχανισμό αυτοαντιστήχησης, όσον αφορά την αξιολόγηση και την κατάρτιση. Άλλε ανησυχίε σχετίζονται με τη χρηματοδότηση και εφαρμογή και υλοποίηση του σώματο ε, αλληλεγγύη σε εθνικό επίπεδο. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα η ετικέτα ποιότητα, πώ δημιουργείται. Δημιουργεί πρόσθετε ε, ευθύνε και ελέγχου για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μια άλλη ανησυχία σχετίζεται με το εξή, ότι η εφαρμογή αυτού του σώματο εξαρτάται από τι υποδομέ του Erasmus Plus και κατά πόσο οι εθνικοί φορεί έχουν επαρκεί πόρου ώστε να πετύχουν όλου του στόχου. Τελική ανησυχία σχετικά με αυτό αφορά την ε, κατανομή της χρηματοδότησης επίπεδο κρατών μελών. Η παρούσα πρόταση, αντίθετα από τον οργανισμό Erasmus Plus, δεν παρέχει κάποια ένδειξη σχετικά με το πώς οι δραστηριότητες και οι προπολογισμοί κατανέμονται μεταξύ κρατών μελών και λήψη συγκεκριμένων πληροφοριών επ' αυτού. Είναι δύσκολο για αυτό το φορέα επί οποία βάσεως συγγνώμη, διανύμονται οι δραστηριότητε αλληλεγγύη στα κράτη-μέλη και πώ οι διάφορε δραστηριότητε λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες κάθε χώρα. Συστήνουμε ότι η πρόταση θα πρέπει να αναφέρεται λεπτομερώς στου στόχου, το πεδίο εφαρμογή και τη διακυβέρνηση του ποιοτικού σέμματο, διότι είναι πολύ ευρύ ο ορισμό των δραστηριοτήτων ελληνικής συμμετοχών των φορέων. Λοιπόν, η εφαρμογή και οι διαδικασίε για την εξασφάλιση τη ποιότητα πρέπει να επανεξεταστούν και υπό το φω του φόρτου εργασία που σχετίζεται με την εξέταση ποιότητα κάθε ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα που θα πρέπει να κινηθεί πόσο θα φορτωθεί από αυτή τη διαδικασία. Η πρόταση θα πρέπει να προβλέπει μηχανισμό για την κατανομή του προπολογισμού στα κράτη-μέλη και οι εθνικοί φορεί για καθήκοντα θα πρέπει να εκτελούν όσον αφορά την εξασφάλιση τη ποιότητα και την υλοποίηση και την υποστήριξη. Τελευταία ομάδα ανησυχιών σχετίζεται με το ελεγκτικό πλαίσιο και μη συμμόρφωση Δηλαδή, το πλαίσιο ελέγχου δεν έχει ακόμα αναπτυχθεί και δημιουργεί ερωτηματικά για το πώ η συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Σώματο Αλληλεγγύη στου γενικού στόχου, ενίσχυση τη συνοχή και την αλληλεγγύη στην Ευρώπη, πώ θα αξιολογηθούν οι στόχοι, αν επιτυχάνονται. Άλλη ανησυχία. Ορισμό των δραστηριοτήτων αλληλεγγύη διευκρινίζει τι απαιτήσει τη πτυχή τη αλληλεγγύη. Πώ καλύπτεται τι δραστηριότητε. Ευρύ ορισμό οδηγεί σε σύγχυση όσον αφορά τα όρια του οργανισμού. Ποιοι φορεί μπορούν να συμμετάσχουν για, ποιο, για την ετικέτα ποιότητα και πώ καλύπτονται οι ανάγκε οι κοινοτικέ. Και πώ μπορούν να ταιριάξουν οι εθελοντέ με τι εργασίε που κάνουν στι ανάγκε τι διάφορε. Τέλο, κατά πόσο αυτή, αυτό το σήμα ποιότητα ε, μπορεί να, να εμποδίσει την κάλυψη θέσεων εργασίας κανονικές από εθελοντισμό. Οι δραστηριότητε αλληλεγγύη μπορούν να ερμηνευθούν ευρέω, οπότε χρειάζεται ανάλυση. Όσον αφορά το σήμα ποιότητα, ούτω ώστε να μην αντικαθίστανται οι θέσει εργασία από θελοντισμό, έχουμε κάποιε συστάσει σχετικά με αυτό. Για να αξιολογήσουμε κατά πόσο η πρόταση αυτή για το σώμα πετυχαίνει του στόχου, η πρόταση πρέπει να εξηγεί καλύτερα το πώ συμβάλλει το σώμα αυτό εθελοντισμού στα προβλεπόμενα αποτελέσματα. Και εκεί συμπεριλαμβάνουμε ότι οι δείκτε που καθορίζονται θα πρέπει να ισχύουν για να ελέγχεται πρώτα απ' όλα η πρόοδο στην επίτευξη του αποτελέσματο και δεύτερον, στο βαθμό στον οποίο συμβάλλει αυτό το σώμα στην επίτευξη των στόχων των άλλων προγραμμάτων που χρηματοδοτούν το σώμα. Η ανάπτυξη ενό πλαισίου παρακολούθηση δεν μπορεί να περιμένει μέχρι 6 μήνε μετά τη θέση ισχύ του κανονισμού. Η νομοθετική πρόταση θα πρέπει να αποσαφηνίζει τι εννοούμε με δράσει δράσεις αλληλεγγύης για τους διάφορους φορείς που συμμετέχουν. Και η πρόταση θα πρέπει να αναφέρει ρητά πώς αποφεύγεται η κατάχρηση και η αντικατάσταση τη αμοιβόμενη εργασίας. Θα, ε, θα έπρεπε να μπει στο Erasmus Συν. Εάν είχε ενταχθεί στο Erasmus Συν, ο κανονισμός θα γινόταν περίπλοκος. Γι' αυτό απερίφθη η ένταξη του σώματος στο Erasmus Plus. Πρέπει να εξεταστούν αυτά τα κριτήρια. Και θα πρέπει να εξηγηθεί καλύτερα αυτή η επιλογή. Όσον αφορά το επιχείρημα του περίπλοκου χαρακτήρα, το Erasmus ε, Plus καλύπτει το 60% του προπολογισμού, παρέχει υποδομέ και οι δράσεις μη κινητικότητας είναι ένα κομμάτι μόνο της, ε, του προγράμματος και είχε χρησιμοποιηθεί αλλιώ το σήμα το ποιοτικό στι διαπραγματεύσει. Το αντίθετο επιχείρημα για να ενταχθούν διάφορα προγράμματα σε ένα, οι δράσει αλληλεγγύη θα μπορούσαν να ωφεληθούν από το σήμα το ποιότητα του Εράσμου. Και ελπίζω ότι αυτή η μελέτη θα τροφοδοτήσει τη συζήτηση για το νομοθέτημα αυτό και θα, τελικά θα συμβάλλει στο να υπάρχει μια ευρωπαϊκή διάσταση στις δράσεις αλληλεγγύης. Yeah, Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίαση της μελέτης σας που θα φανεί πολύ χρήσιμη στο από εδώ και πέρα έργο μας, ιδίως όσον αφορά τις, τα αιτήματα που, στα οποία καταλήξατε, στις απαιτήσει που καταλήξατε, τις οποίες ενδεχομένως χρειάζεται να εντάξουμε με έναν πιο συγκεκριμένο τρόπο και στην έκθεση που θα συντάξουμε. Και τώρα περνάμε στην οπτική των εθνικών φορέων, των εθνικών ε, υπηρεσιών, Καλωσορίζω λοιπόν για άλλη μια φορά τον κύριο Μάνφρετ Φον Χέμπελ και του δίνω το λόγο για πέντε λεπτά. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που μα δίνετε τη δυνατότητα να συμβάλλουμε στην συζήτηση. Το δίκτυο των εθνικών φορέων υποστηρίζει βεβαίω το στόχο και την ιδέα τη δημιουργία ενό Ευρωπαϊκού σώματο αλληλεγγύη. Είναι ε, ένα εργαλείο που είναι απαραίτητο για την ενίσχυση τη κοινωνική συνοχή και τη αλληλεγγύη στην Ευρώπη. Ταυτόχρονα το σώμα αυτό ε, θα βοηθήσει στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας και στην απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων. Θεωρούμε ότι βασική εστίαση του σώματος θα πρέπει να είναι η δημιουργία μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας και της ιδιότητας του ενεργού Ευρωπαίου πολίτη. Η κοινωνική συνεχή και η ελεγγύη βεβαίω δεν μπορεί να προέλθει απλά με την υλοποίηση ενό προγράμματο. Χρειάζεται να μάθουμε και να παρακολουθήσουμε, να αφουγκραστούμε ποιε είναι οι εμπειρίε των νέων ανθρώπων που θα συμμετάσχουν σε αυτό το σώμα. Πρέπει λοιπόν το, το μήνυμα ε, να είναι σαφέ ότι θα υπάρχει μια έντονη ευρωπαϊκή διάσταση στο σώμα αλληλεγγύη. Ιδίω όσον αφορά τα προγράμματα και τα έργα που θα υλοποιούνται εντό μια χώρα που δεν έχουν από φυσικού τους μια τέτοια ευρωπαϊκή διάσταση, απαραίτητος τουλάχιστον. Μια από τις βασικές μας ανησυχίες αυτή τη στιγμή είναι ο περιορισμός του γεωγραφικού πεδίου ισχύου του σώματος. Εμείς πιστεύουμε Έτσι λοιπόν φαίνεται αυτό ε, ε, στην πρόταση ότι αυτό το σήμα είναι πολύ απογοητευτικό για τις χώρες που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών, τις υποψήφιες αλλά και τις χώρες εταίρους νομίζω ότι πρέπει να εξασφαλιστεί με κάθε ε, τρόπο η συμμετοχή όλων των χωρών και πρέπει επίσης να φροντίσουμε ώστε το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης να συμπεριλαμβάνει και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθερών Συναλλαγών από την αρχή μάλιστα, από την φάση της εκκίνησης του προγράμματος αυτού. Επίσης, νομίζω ότι πρέπει να καταστεί δυνατή και η συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου έως το τέλος του προγράμματος. 2020, λέει ο μιλητής, απαντώντας σε κάποια ερώτηση την οποία δεν ακούσαμε όμως. Αναφέρθηκε η κοινωνική ένταξη, η πυκλομορφία, η διαφορετικότητα. Κανείς δεν πρέπει, κανένας νέος άνθρωπος δεν πρέπει να, να αντιμετωπίσει φραγμούς και εμπόδια ως, την, ε, ως προς την πρόσβαση του σε αυτό το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Ωστόσο κάποιοι άνθρωποι με ειδικές ανάγκες ή που έχουν λιγότερες ευκαιρίες χρειάζονται ε, συγκεκριμένη υποστήριξη και θα πρέπει αυτή η διάσταση να τύχει ιδιαίτερη εστίαση και προτεραιότητα στο πρόγραμμα. Χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερη υποστήριξη και αρρωγή στους νέους ανθρώπους ε, που ανήκουν σε μειονεκτούσες πληθυσμιακές ομάδες. Πολλές φορές αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται εκτός οργανώσεων, δεν συμμετέχουν στην κοινωνική ζωή, γι' αυτό και χρειάζεται ε, επαρκής χρηματοδότηση και υποστήριξη προκειμένου να μπορέσουμε να φτάσουμε και σε αυτούς τους ανθρώπους ε, και στις οργανώσεις που ενδεχομένως έχουν στο επίκεντρο της προσοχής τους αυτές τις πληθυσμιακές ομάδες. Όπω έχει αναφερθεί ήδη αρκετέ φορέ, στο πλαίσιο του προτινούμενου κανονισμού, η διαφορά ανάμεσα στον εθελοντισμό, τι πρακτικέ ασκήσει και τις θέσει εργασία δεν είναι επαρκώ σαφής. Όπως είπε πολύ σωστά και ο Σάιμον ε, και όπω προκύπτει από τη μελέτη, και εμείς ε, θεωρούμε ότι υπάρχει μια θολότητα όσον αφορά την ε, συμμετοχή των διαφόρων ε, ομάδων στο πρόγραμμα, αυτό μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην πορεία. Χρειαζόμαστε ξεκάθαρους ορισμούς για κάθε τομέα, χρειαζόμαστε καλύτερες περιγραφές ε, των μορφών ε, και των τύπων των προσφερόμενων υπηρεσιών, του εθελοντισμού, των πρακτικών ασκήσεων, των θέσεων εργασίας. Θεωρούμε ότι χρειάζεται αυτή η ευρωπαϊκή διάσταση να διακριθεί και από το γεγονός ότι δεν θα υποκατασταθούν ε, ε, θέσεις απασχόλησης πραγματικές μέσω ε, δραστηριοτήτων αλληλεγγύης. Επίσης, θεωρούμε ότι οι ιδιώτες θα πρέπει να μπορούν μεν να συμμετέχουν αλλά μόνο εφόσον έχουν μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Υπάρχει ένα υψηλό πρότυπο ποιότητας όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Σώμα, την, την Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία και νομίζω ότι αυτό το υψηλό πρότυπο πρέπει να διατηρηθεί και στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Αναφέρομαι στην κατάρτιση, στην κατάρτιση στους κύκλους εκπαίδευσης, υπάρχουν όλα αυτά ε, που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Άρα ξεκινάμε από μια πολύ θετική βάση. Υπάρχει ήδη μια πολύ σημαντική ε, βάση ανθρώπων που συμμετέχουν με εξασφάλιση υψηλών προδιαγραφών ποιότητας σε, το, στις υπάρχουσες υπηρεσίες και νομίζω ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε ε, τη βάση του προγράμματος που θα πρέπει να είναι οι συμμετέχοντες σε συνεργασία με τις εθνικές υπηρεσίες αλλά και τις συμμετέχουσες οργανώσεις. Νομίζω ότι πρέπει να διατηρηθεί το Youth Pass ε, ως ε, διαπιστευτήριο για να συμμετάσχει κανείς σε αυτόν. 700.000 πιστοποιητικά έχουν ήδη διανεμηθεί ε, για συμμετέχοντες ε, σε δράσεις για την νεολαία και νομίζω ότι είναι ένα εργαλείο που αποδείχθηκε πολύ σημαντικό και πολύ χρήσιμο. Τέλος, ε, η αλλαγή του, του, του πόρταλ του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης ε, είναι απαραίτητη, διότι αυτή τη στιγμή δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των συμμετεχόντων και των οργανώσεων. Αυτή τη στιγμή αποτελεί μια καλή βάση, μια καλή μαγιά, αλλά όταν περάσουμε στην πραγματική εφαρμογή του προγράμματος, νομίζω ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη πολύ περισσότερο και πολύ, ε, σε πολύ, με πολύ σοβαρότερο τρόπο οι ανάγκες ε, και οι επιθυμίες των ίδιων των συμμετεχόντων και των οργανώσεων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το δίκτυο εθνικών φορέων βεβαίως έχει ε, παράσχει ε, πολύ λεπτομερέστερες ε, ε, παρατηρήσεις και σχόλια στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και είμαστε στη διάθεσή σας όποτε μας χρειαστείτε. Ευχαριστώ λέει η Πρόεδρος. Ήμουν αρκετά γενναιόδορη με το χρόνο που σας έδωσα. Σας ευχαριστώ για την συμβολή σας αυτή στη συζήτηση και περνάμε στον Πρόεδρο Πάβελ Τραντίνα πρόεδρο του Τμήματος ε, Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόλησης ε, που θα μας παρουσιάσει τη γνωμοδότηση που συνέταξε η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Έχετε τρία λεπτά κύριε Γαντίνα, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε που μου δίνετε την ευκαιρία να σας ε, παρουσιάσω την γνωμοδότηση των εργοδοτών, των συνδικάτων και άλλων ε, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που εκπροσωπούνται στην Επιτροπή ε, Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σχέδιο γνωμοδότησής μας εγκρίθηκε ομόφωνα από το δικό μου τμήμα. Τώρα θα πρέπει πια να εγκριθεί επισήμως από την Ολομέλειά μας την επόμενη εβδομάδα, πράγμα που ελπίζουμε ότι θα γίνει χωρίς σημαντικές αλλαγές. Σε σχέση με την Οικονομική και, η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ορίζει την ε, πρόταση της Επιτροπής και θεωρεί ότι είναι καλό σημείο κίνησης για περαιτέρω συζήτηση, αλλά πιστεύουμε πως πρέπει πολλά στοιχεία να διευκρινιστούν. Ήδη ακούσαμε διάφορες παρατηρήσεις από ε, τους προλαλήσαντες. Θα ξεκινήσω με την πρώτη μου παρατήρηση και αυτό είναι το θέμα το οικονομικό. Ανησυχούμε ότι αυτή η νέα επένδυση στον εθελοντισμό, στους νέους και στην αλληλεγγύη θα επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό μέσω της ανακατανομής χρημάτων από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εθελοντισμού. Και αυτή η επένδυση νομίζουμε πως δεν θα πρέπει να γίνει εις βάρος επιτυχών προγραμμάτων που ήδη προσφέρουν πολύτιμες ευκαιρίες στους ε, νέους και κυρίως στο Erasmus Plus που ήδη ε, υποχρηματοδοτείται όπως γνωρίζουμε και μάλιστα ε, το Εράσμου θα έπρεπε κανονικά να παραπλασιαστεί επί 10 και ξεκινάμε μια τέτοια εκστρατεία. Και αυτό σημαίνει ότι θα έπρεπε να έχουμε φρέσκο χρήμα γι' αυτό εδώ το πρόγραμμα. Επίσης ε, μας ανησυχεί πολύ η συγχώνευση των στόχων του σώματος αλληλεγγύης με αυτό των πολιτικών για την απασχόληση των νέων. Γι' αυτό και η Επιτροπή μας προτείνει μετά από αίτημα των κοινωνικών εταίρων μάλιστα η συμπερίληψη των μαθητιών και των θέσεων απασχόλησης να επανεξεταστεί. Καλύτερα θα ήταν να ενδυναμωθούν αυτά τα στοιχεία στα υπάρχοντα προγράμματα, εστιάζοντας στην απασχόληση και τις μαθητείες και όχι σε αυτό το νέο πρόγραμμα. Και επίση, ε, υπάρχουν πλονεκτήματα εάν συγκεντρωθούν μόνο στον εθελοντισμό αυτό το σώμα θα σημάνει μεγαλύτερη σαφήνεια, εστιασμό και θα απεφευθεί η σύγχυση με άλλα προγράμματα για τους νέους που υπάρχουν για την υποστήριξη της απασχόλησης των νέων. Μετά από ευρείες ε, διαβουλεύσεις με βασικούς ε, ενδιαφερόμενους φορείς, η Επιτροπή μας ε, έχει να κάνει άλλες προτάσεις για τη βελτίωση του σχεδίου κανονισμού. Ήδη θα έχετε λάβει το σχέδιο γνωμοδότησης, αλλά να τονίσω κάποια στοιχεία. Ο ορισμός των, των δράσεων εθελοντισμού θα πρέπει να αποσαφενιστεί. Το, επίσης η θύρα θα πρέπει να είναι ένα πραγματικό μέσο interacti, ε, ε αλληλεπίδρασης, δράσης και διάδρασης, δηλαδή διπλή και αμφίδρομη ε, ε, δυνατότητα δραστηριοποίησης και των νέων και της διοίκησης. Οι οργανώσεις των νέων θα πρέπει να προετοιμάζουν ε, τους νέους με ε, ειδικέ ανάγκες για να συμμετέχουν στον εθελοντισμό. Θα πρέπει επίσης ε, το, η βασική διαχείριση να γίνεται από την Κομισιόν να αυξηθεί η, η δυνατότητα πρόσβασης όπως και η εθνικοί φορείς να αλλάξουν ώστε να είναι πιο φιλικοί προς το χρήστη. Κάτι ακόμα έχει να κάνει με το πού θα πρέπει να βρίσκεται το σώμα αλληλεγγύης. Θα πρέπει να μείνει μέσα στο υφιστάμενο πρόγραμμα Εράσμος ΣΥΝ αντί να δημιουργηθεί ένα τελείως νέο πρόγραμμα, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αυτό θα συνδυάσει τους όρους του, του, του, του υπολείπου της ε, εθελοντικής υπηρεσίας με το σώμα αλληλεγγύης. Γιατί διαφορετικά θα έχουμε δύο παρόμοια προγράμματα που θα έχουν όμως ε, έδρα γεωγραφική αλλού. Και το Erasmus Plus και το Σώμα Αλληλεγγύης δεν θα απειληθούν ε, μετά το 2020. Πολύ ανησυχούμε γι' αυτό. Ε, εν πάση περιπτώσει χρειάζεται επιπλέον χρηματοδότηση και στήριξη να κλείσω με κάτι το ευρύτερο. και αυτό αφορά τις ε, πολιτικές ε, εθελοντισμού. Ελπίζουμε ότι μέσω αυτού του προγράμματος ε, θα υπάρξει και θα σχηματιστεί μια ευρύτερη ευρωπαϊκή πολιτική για τον εθελοντισμό, όχι μόνο για τους 100.000 εθελοντές, αλλά για, περίπου, για το περίπου ένα εκατομμύριο νέους και, και λιγότερο νέους εθελοντές, ευρωπαίους πολίτες που αυτή τη στιγμή ε, συμμετέχουν σε εθελοντικά προγράμματα. Όπω ήδη έχουμε τονίσει στη γνωμοδότησή μας τη ΟΚΕ για τις εθελοντικέ πολιτικές και την Ένωση το 2011, πιο συντονισμένη προσέγγιση χρειάζεται από πλευράς όλων των ευρωπαϊκών θεσμών όσον αφορά τις εθελοντικές ε, πολιτικές. Θα πρέπει να θεωρηθεί μια οριζόντια πολιτική και να, ε, να, να προωθηθεί από τις δομές των ευρωπαϊκών θεσμών. Και προς αυτό θα ήθελα να σας θυμίσω αυτή τη δημοσίευση που μπορεί να θυμάστε ότι την κάναμε το 2011. Η συντάκτρια, μία εκ των συντακτριών βρίσκεται εδώ δίπλα μου. Γύρω στους 100 ειδικού εργάστηκαν από αυτής. Είναι η ατζέντα πολιτικής για τον εθελοντισμό. Μπορεί να προσφέρει πολλά ε, στοιχεία έμπνευσης για τον κανονισμό. Ευχαριστώ πολύ. Και Περνάμε τώρα στην ε, Γκαμπριέλα Σίβικο που είναι διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Εθελοντισμού. Έχετε το λόγο για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι είναι ευπρόσδεκτη αυτή η προσοχή που δίνεται στην αλληλεγγύη και στον θελοντισμό. Πρέπει να απαντηθούν όμως κάποιες ερωτήσεις όπως είπαν και οι Δηλαδή, περί τίνο πρόκειται. Τι εννοούμε με το σώμα αλληλεγγύη, γιατί το χρειαζόμαστε και πώς θα το διαχειριστούμε. Περί τίνο πρόκειται. Γιατί πράγμα μιλάμε. Μιλάμε για αλληλεγγύη. Ελπίζουμε ότι όλες οι δράσεις θα εμπνέονται από την αλληλεγγύη προς τους άλλους. Θα πρέπει διάφοροι φορεί που έχουν βασικό σκοπό να παράξουν εισόδημα για τους μετόχους τους, αυτού του είδου οι φορεί θα πρέπει να φιλοξενούν συμμετέχοντες στο σώμα αλληλεγγύης, αν γίνεται αυτό, θα είναι ασύμβατο. Άρα οι ε, κερδοσκοπικοί φορείς θα πρέπει να αποκλειστούν. Αν θέλουν να συμμετάσχουν με τα χαράς, ε, θα το ενθαρρύνουμε, οι κερδοσκοπικές επιχειρήσεις να δημιουργήσουν συμπράξεις με μη κυβερνητικές οργανώσεις, κοινωνία των πολιτών και διάφορους άλλους φορείς, αλλά δεν θα πρέπει άμεσα να συμμετέχουμε Όπως είπαν και άλλοι Χρειάζεται σαφής διάκριση μεταξύ μαθητείας, θέσεων απασχόληση και θελοντισμού. Πρέπει να λάβουμε υπόψη τα πολλαπλά νομικά πλαίσια που καλύπτουν τι διάφορε προσεγγίσεις στην Ευρώπη. Και αυτή η νομική πρόταση ε, δεν το καταφέρνει ακόμα. Λοιπόν, οι σκοποί του εθελοντισμού και της μαθητείας πρέπει να σαφώνονται. Ο εθελοντισμός έχει στόχο την κάλυψη αναγκών, κοινωνικών αναγκών. Εκφράζει αλληλεγγύη. Και δευτερεύον παράγον είναι αυτά που μαθαίνει ο εθελοντής. Στη μαθητεία, για μια ποιοτική μαθητεία, πρωτίστως στόχος είναι η εκμάθηση ε, διαφόρων γνώσεων από πλευρά του μαθητευόμενου. Κάτι άλλο που μα ανησυχεί είναι ότι σταζόμεθα εδώ επί αυτοαπασχόλησης ή επιχειρηματικότητας. Η ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων είναι πασίγνωστο φαινόμενο όταν κανείς συμμετέχει στον θελοντισμό, αλλά επουδενή θεωρούμε ότι θα πρέπει να ενθαρρύνουμε ανθρώπου να συμμετέχουν σε εθελοντικέ δράσει, ούτω ώστε να κερδίσουν προσωπικά κέρδη, να αποκομίσουν κέρδη από αυτή την εμπειρία. Και προτείνουν συγκεκριμένη τροπολογία για να αποφευθεί σύγχυση. Δηλαδή ότι οι νέοι θα συμμετέχουν σε δραστηριότητε αλληλεγγύη, ούτω ώστε να αποκτήσουν κέρδη προσωπικά και οικονομικά στο τέλο τη διαδικασία. Γιατί χρειαζόμαστε το σώμα αλληλεγγύη. Του τελευταίου μήνε πολύ διαρωτηθήκαμε. Εάν υπάρξει αν καρποφορήσει αυτή η προσπάθεια, θα πρέπει να συμπληρώνει τι ισχύουσε πρωτοβουλίε και να δίνει προστιθέμενη αξία. Και η πρόταση ω έχει δεν αναγνωρίζει επαρκώ τα πολλά εκατομμύρια θελοντών και εκατοντάδες χιλιάδες οργανισμού και φορεί που ήδη παρέχουν δραστηριότητε πολύ ποιοτικέ αλληλεγγύη. και αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στο πρόγραμμα. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης έχει δυνατότητες. Μπορεί να είναι μια πύλη για μια διαβίου ε, εθελοντική δράση και θα δίνει τη δυνατότητα να ενισχυθούν οι οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών με ανθρώπινους πόρους που χρειάζονται διακαώς, κυρίως λόγω των μέτρων λιτότητας δημιουργείται αυτή η ανάγκη, για να μπορέσουν να κάνουν σωστή επιλογή εάν δέχονται ανθρώπους για μαθητή αυτή οι ή θα προσλαμβάνουν κάποιο θελοντή, κάθε τοποθέτηση θα πρέπει να αμείβεται ισότιμα, να χρηματοδοτείται ισότιμα. Χρηματοδοτούνται πλήρως μόνο οι θέσεις εθελοντισμού και οι θέσεις μαθητές όχι. Άρα κάποιος μπορεί να κάνει λάθος επιλογή. Όταν μια τοποθέτηση θα αποκαλύπτει, θα αποκαλύπτε ότι μια θέση εθελοντική ενώ βασικά θα είναι θέση μαθητείας. Διαχείριση του προγράμματος. Συμμετοχή των διαφόρων φορέων πρέπει να αναγνωριστούν επαρκώς όλα τα υφιστάμενα δίκτυα, φορείς εθελοντισμού, φορείς ε, δικτύωσης των νέων, εκπροσώπησης των νέων, ε, όσοι ε, θα συμμετέχουν στην εφαρμογή υλοποίηση του προγραμμάτου Το, το κέντρο πόρων του ευρωπαϊκού σώματος εθελοντισμού θα πρέπει να κατατεθεί μέσω ανοιχτού διαγωνισμού να μην ανατεθεί στους φορείς του Erasmus Plus αυτόματα. Χρειάζεται ένα ευρύτερο φάσμα φορέων και οργανισμών να συμμετέχουν με τεχνογνωσία όσον αφορά τον των νέων, αλληλεγγύη των νέων, απασχόληση των νέων και ενημέρωση των νέων. Όλοι αυτοί να συμμετέχουν στην πρωτοβουλία. Όπω είπαν και οι προλαλήσαντε, χρειάζεται μεγαλύτερη σαφάνεια όσον αφορά τι έννοιε και του ορισμού. Ευπρόσδεκτε οι μορφέ των διαφόρων φορέων ε, και των διαφόρων τοποθετήσεων θα πρέπει ε, να είναι ξεκάθαρο οπότε υπάρχει εθελοντική συμμετοχή. Έχουμε πιο λεπτομερή ανάλυση στη μακροσκελή έκθεση. Εάν θέλουμε να έχουμε και τους δύο κλάδους εθελοντισμού και μαθητείας πρέπει να γίνεται σαφής διάκριση ε, εμπειρία Ευρώπη, κάτι που δίνει δυνατότητα στους νέους Φερρυπίν να αυξήσουν την απασχολησιμότητά τους, είναι ένας κλάδος και σε άλλο κλάδο ξεχωριστό να δίνουμε τη δυνατότητα στους νέους να εκφράζουν αλληλεγγύη. Ο Πάβελ ήδη είπε αυτό που θέλω να πω στο τέλος. Όλα αυτά θα πρέπει να ενταχθούν σε μια πλήρη στατηγική εθελοντισμού. Δεν πρέπει να είναι μια μεμονωμένη ε, πρωτοβουλία, θα το στηρίξουμε αυτό. Θέλουμε να δημιουργηθεί μια πραγματικά, ένας πραγματικός, μια κουλτούρα εθελοντισμού στην Ευρώπη. Ευχαριστούμε πολύ. Και περνάμε τώρα στο γύρο ερωταπαντήσεων. Θα ήθελα να δώσω το λόγο πρώτα στους σκιώδεις εισηγητέ των δύο επιτροπών, εφόσον βεβαίως επιθυμούν να λάβουν το λόγο. Σας παρακαλώ μόνο ερωτήσεις και όχι περισσότερο από ένα λεπτό. Ο κύριος Κλούνεφ. Η κυρία Κλούνεφ. Συγγνώμη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για όλες αυτές τις παρουσιάσεις. Νομίζω ότι ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που ακούσαμε. Αυτό που ε, κρατάω εγώ ως σήμα και ως μήνυμα είναι ότι δεν πρέπει να υπάρξει σύγχυση ανάμεσα στον εθελοντισμό και την πρακτική άσκηση, τις μαθητείες. Εγώ αναγνωρίζω την αξία του εθελοντισμού και θεωρώ ότι μπορεί να ενισχύσει με εμπειρίες το άτομο, ε, εμπειρίες που θα αποκομίσει και τις οποίες μπορεί να αξιοποιήσει και στην πορεία της ζωής του ε, σε τέτοιου είδους προγράμματα με κοινωνικό χαρακτήρα, κάτι που δεν θα συνέβαινε απαραίτητα με μια απλή θέση απασχόλησης. Απλά, θα ήθελα να ρωτήσω τον Επίτροπο άλλη μια φορά όσον αφορά την χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση θα προέλθει από τα διάθετα κονδύλια του προγράμματος Εράσμους. Κατάλαβα σωστά. Γιατί κάποια μέλη ε, έθεσαν ε, το ζήτημα ότι υπάρχει ανάγκη να εξευρεθεί νέα, φρέσκια χρηματοδότηση. Η κυρία Τσόντροβα από την Επιτροπή Πολιτισμού έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους εμπειρογνώμονες που έλαβαν το λόγο. Εγώ λοιπόν διαπίστωσα ότι υπάρχει ένα νήμα που διατρέχει όλες τις τοποθετήσεις που ακούσαμε. Ότι οι στόχοι του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης θα πρέπει να αποσαφινιστούν. Να ξεκαθαριστεί δηλαδή ποιος θα είναι ο ρόλος που θα διαδραματίσει αυτό το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, ποιος θα είναι ο ρόλος των πρακτικών ασκήσεων των μαθητιών. Ε, νομίζω ότι αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου να στεφθεί η όλη πρωτοβουλία με επιτυχία. Ένα ακόμη ερώτημα. Ο Επίτροπος είπε σαφώς ότι το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα συμπεριλαμβάνει όλες τις δράσεις αλληλεγγύης. Αυτό σημαίνει ότι θα συμπεριλαμβάνει και τις υφιστάμενες δράσεις και θα τις καλύπτει αυτές. Αυτό σημαίνει ότι οι άλλες δραστηριότητες, οι άλλες δράσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη με κάποιον τρόπο δηλαδή θα μεταφερθούν στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και μιλώ συγκεκριμένα για την Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία που έχει και εκείνη μια έντονη διάσταση αλληλεγγύης. Θα υπάρχει ε, αυτόνομη από εδώ και πέρα πορεία αυτή τη Ευρωπαϊκή Εθελλοτική Υπηρεσία ε, στο σώμα ηλελλήσει. Η κυρία Σίλβια Κώστα έχει το λόγο. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ δεν κατάλαβα καλά στο σωμα αλληλεγγυη η κυρια σιλβια κωστα εχει το λογο ευχαριστω προεδρε εγω δεν καταλαβα καλα στο τελος αν εσείς θεωρείτε πως... Ε, σε σχέση με τη βασική διάκριση ανάμεσα στην εργασία και τον εθελοντισμό αν αυτό σημαίνει και αποδοχή ή όχι των ιδιωτικών εταιριών και όχι μόνο των non-profit. στην κοινωνική οικονομία των συμμετεχόντων ή νομίζετε ότι αρκεί να γίνει αυτή η διάκριση στο κείμενο γιατί κατά τη γνώμη μου αυτό προέκυψε και από τις υπόλοιπες παρεμβάσεις, ότι δηλαδή μπορεί να δημιουργηθεί μια γκρίζα αγορά, δηλαδή όχι μόνο εργασία που παίρνει τη μορφή εθελοντισμού, αλλά και ο ίδιος ο εθελοντής να μην μπορεί να αμυφθεί αργότερα για την ε, αμοιβόμενη εργασία, την οποία ωστόσο κάνει. Τώρα, εδώ για σας Επίτροπε. Μιλάμε για χώρες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ από την αρχή θεωρώ πως θα ήταν σημαντικό να μην ε, σταματήσει η προσοχή που δίνεται σε τρίτες χώρες που ήδη συμμετέχουν ας πούμε στο Εράσμος. Είναι 33 οι χώρες και τις τρίτες χώρες. Επίσης, κάτι ακόμα. Υπάρχουν άλλοι δύο κίνδυνοι. Θα τις συζητήσουμε ίσως αργότερα και προέκυψαν και στη συζήτηση. Το ένα είναι το θέμα της ευρωπαϊκής προστιθέμενης Αξία, που κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να υπάρχει πάντα ακόμα και όταν είναι μέσα σε μία μόνο χώρα, να είναι δηλαδή παιδιά από διάφορες εθνικότητες. Και έπειτα η επικάλυψη με τα εθνικά συστήματα. Εδώ λοιπόν βλέπω εγώ τα προβλήματα και ήθελα και περαιτέρω διευκρινήσεις. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Κούρτσιο Μαλτέζε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ συμμερίζομαι τι παρατηρήσει όσον αφορά τη διάκριση ανάμεσα στην εργασία και την αλληλεγγύη, γι' αυτό δεν θα το συζητήσω εδώ, αλλά θέλω να κάνω μια ερώτηση στον Επίτροπο Ναύρατζιτ. Ξέρουμε πως υπάρχουν προγράμματα όπω το Erasmus Plus που θα χρειαζόταν περισσότερη χρηματοδότηση και είναι άδικο να αφαιρείται χρηματοδότηση για άλλε πρωτοβουλίε από αυτό. Γνωρίζουμε όμως και ότι υπάρχουν πολύ ισχυρές αντιστάσεις πολιτικές να δημιουργηθούν νέε μορφέ χρηματοδότησης. Όμω υπάρχουν και προγράμματα που δεν απορροφούν τελείω το μπάτζετ του, ας πούμε το Ταμείο αλληλεγγύη. Διερωτώ με και σας ρωτώ, δεν είναι δυνατόν με κάποιο τρόπο εφόσον δεν έχουν απορροφηθεί όλα αυτά τα κονδύλια, να χρησιμοποιήσουμε το Ταμείο Αλληλεγγύης, που ναι, είναι θέμα, ε, ε, ε, είναι κονδύλια που αντιμετωπίζουν επίγουσες ενάγκες αλλά θα μπορούσε να λειτουργήσει και ως πρόληψη, περιμένοντας να βρούμε την πολιτική συνένεση για να αυξηθεί η χρηματοδότηση στις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες αλληλεγγύης. Ευχαριστούμε και μιας και έχετε με δύο ιδιότητες σήμερα εδώ, ε, δεν σας έλαβα υπόψη μου. Ε, νόμιζα ότι ήσασταν ο εισηγητής της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. Όμως βλέπω ότι είστε και μέλος της, Ευρω... της Επιτροπής Απασχόλησης. Κύριε Ρέγμαν, κύριε Ρέγμαν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δύο σχόλια έχω. Κύριε Επίτροπε, κυρίε και κύριοι. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά την πρόταση για 80% εθελοντική δράση και 20% ε, κατάρτιση ή απασχόληση. Όσον αφορά αυτό τον επιμερισμό, θα ήμουν αντίθετος. Πρέπει το ποσοστό απασχόλησης να ε, αυξηθεί εις βάρος του εθελοντισμού. Η εθελοντική δράση είναι πάρα πολύ σημαντική. Αλλά Υποτίθεται ότι θέλουμε να βοηθήσουμε την νεολαία, διότι έχει πολύ υψηλά ποσοστά ανεργίας. Και αν θέλουμε να βοηθήσουμε τους νέους, πραγματικά, πρέπει να στείλουμε ένα πραγματικό μήνυμα, σαφές μήνυμα, ότι κάθε νέα θέση απασχόλησης για τους νέους είναι κάτι που ε, επιθυμούμε και μας αφορά. Γι' αυτό προτείνω να έχουμε συνδυασμό 70% εθελοντική δράση και 30% ε, για την απασχόληση. Δεύτερο σχόλιο. Αν το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης έχει στόχο να αντιδρά σε ζητήματα που αφορούν ανοικοδόμηση από καταστροφές, από φυσικές καταστροφές που συμβαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως επί παραδείγματι οι σεισμοί στην Ιταλία ή οι έντονες καταιγίδε στην Πολωνία που έγιναν το καλοκαίρι, ε, Θεωρητικά υπάρχουν ήδη τέτοια συστήματα που λειτουργούν. Είχαμε το παλιό σύστημα εθελοντικής δράσης, ευρωπαϊκής εθελοντικής δράσης. Ξέρετε πόσος καιρός χρειάζεται από όταν υποβληθεί η αίτηση μέχρι να φτάσει κανείς στην τοποθεσία. Ένα εξάμεινο. Κρατάει πολύ. Δεν λέω ότι οι εθελοντές αντικαθιστούν τις τοπικές υπηρεσίες παροχής βοηθείας, αλλά θα έπρεπε να πηγαίνουν σε μια τοποθεσία εθελοντές πιο γρήγορα. Θα ήθελα να επενέσω κατά τα άλλα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έξοχη πρωτοβουλία και την ταχύτητα με την οποία παρουσιάστηκε. Ευχαριστώ. Ο κύριο Ζαριανόπουλο έχει ζητήσει το λόγο ω τελευταίο ομιλητή. Παρακαλώ. Πριν τι ερωτήσει, μια εισαγωγική παρατήρηση που τη βγάζω από την ε, αιτιολογική έκθεση. Ήδη από την πρώτη φράση της αιτιολογικής έκθεσης για το σώμα εθελοντών φαίνεται ότι πρόκειται για μια ακόμη υποκρισία είναι δυνατόν να μιλάς σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση για αλληλεγγύη. Με πολέμους, με επεμβάσεις, με πολλαπλασιασμό των φτωχών, από τους οποίους συνέχεια κόβονται ακόμη και τα ελάχιστα. Για να πάμε όμως και στο συγκεκριμένο ε, ζήτημα και έτσι όπως πολύ παραστατικά δόθηκε και από τις εμπειρογνώμενες εικόνα. Νομίζω ότι η γενική εικόνα είναι ότι υπάρχει μια θολούρα και όσον αφορά τα κονδύλια, την προέλευσή τους, το ύψος τους, αλλά πολύ περισσότερο, και εδώ παίρνω υπόψη μου πολύ και τις δικές τους ανησυχίες, για το μεγάλο γεγονός ότι εδώ μιλάμε πλέον για μια προσπάθεια αντικατάστασης μόνιμης απασχόλησης από ευέλικτη απασχόληση μέσω και αυτού ακόμα του προγράμματος. Ανησυχία που διατυπώθηκε από τους εμπειρογνώμονες. Ανησυχία, ε, όπως, ε, ε, ανησυχία για το είδος των δράσεων. Ποιες θα είναι αυτές για παράδειγμα φυσικές καταστροφές. Στις φυσικές καταστροφές η Ευρωπαϊκή Ένωση την υποστήριξη των χωρών που δέχονται φυσικές καταστροφές δεν τη θεωρεί επιλέξιμη δραστηριότητα. Ενώ κανονικά θα έπαιρνε και να είναι επιλέξιμη αλλά και να υπάρχουν κρατικέ δομέ οι οποίε πραγματικά να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τι ανάγκε των ανθρώπων που δέχονται πλημμύρε, σεισμού ή οτιδήποτε άλλο. Και αυτό κάτι τέτοιο δεν γίνεται. Ή από την άλλη το να υποστηριχθούν άτομα με ανάγκε, ιδιαίτερα φτωχά άτομα κτλ. Πράγμα το οποίο δεν γίνεται. Άρα λοιπόν τελειώνω με αυτό κύριε Πρόεδρε, εδώ μιλάμε πλέον για ένα χάπι εντό εισαγωγικών στην ενεργεία, για μια εκπαίδευση στην ε, ευέλικτη απασχόληση και βεβαίω ξανά για εμπλοκή μη κυβερνητικών οργανώσεων και ιδιωτών που και πάλι θα βγάλουν αρκετά κονδύλια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα να ρωτήσω την εισηγήτριά μα αν έχει ερωτήσει ή παρατηρήσει να κάνει. Ναι. Ήταν πολύ ενδιαφέρον πολύ ενδιαφέρουσα η εμπειρία αυτής της συζήτησης διότι το Τμήμα Πολιτικής μας προφανώς και έχει διαπιστώσει το υψηλό επίπεδο ποιότητας του εθελοντισμού και των δράσεων ε, αλληλεγγύης και ότι ε, δικός, ε, βασικός στόχος πρέπει να είναι η δημιουργία ευρωπαϊκής ταυτότητας. Εγώ νομίζω ότι όσον αφορά το, το γεωγραφικό πεδίο ε, ισχύω πράγματι πρέπει να διευρυνθεί το πεδίο αυτό στα, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών. Ε, νομίζω ότι όσον αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο ε, πρέπει να εξάγει τα συμπεράσματά του και πρέπει και να υποστεί και τις ε, ε, επιπτώσεις των αποφάσεών του. Ε, Erasmus πλάς και δεκαπλασιασμός της χρηματοδότησης. Βεβαίως ήταν πάρα πολύ, θα ήταν πάρα πολύ ωραίο κάτι τέτοιο. Όπως είπε και ο Παύλ Τραντίνα, πράγματι δεν πρέπει να υπάρξει σύγχυση ανάμεσα στην εργασία και στον εθελοντισμό και ε, όσον αφορά την αύξηση των χρηματο... της χρηματοδότησης για το Erasmus Plus έως το 2020 ε, εγώ θεωρώ ότι δεν είναι απαραίτητο Sony και δεν, δηλαδή να ενταχθεί το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης ε, στο Erasmus Plus ενδεχομένως και μια λύση δύο αυτόνομων προγραμμάτων να έχει και εκείνη τα πλεονεκτήματα της. Επίσης, όπως είπε η κυρία Σίβικο, πιστεύω και εγώ ότι όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να κινητοποιούνται και να παροτρύνονται από ένα εσωτερικό αίσθημα αλληλεγγύης και όχι από ιδιωτελείς σκοπούς. Νομίζω επίσης ότι τα προγράμματα θα πρέπει να έχουν ε, ρίζες κάτω στη, βάση, στις ε, τοπικές κοινωνίες και ε, μου έκανε εντύπωση βεβαίως πρέπει να σημειώσω το γεγονός ότι ε, πολλοί εκπρόσωποι των δεξιών κομμάτων ε, θεωρούν ότι δεν πρέπει να ενισχυθεί η, ότι, η αλληλεγγύη ενώ από την άλλη ακούσαμε τον Έλληνα κομμουνιστή να μας λέει ότι ε, δεν υπάρχει καμία ε, αλληλεγγύη στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να δώσω την ευκαιρία στους εμπειρογνώμονες μας να απαντήσουν σε όποιες ερωτήσεις θεωρούν εκείνοι ότι ε, αξίζει να απαντήσουν ή μπορούν να απαντήσουν. Γιατί ε, είμαστε κάπως, έχουμε κάποιον χρονικό περιορισμό πρέπει να σας πω. Κύριε Μπρούκ. Δεν μου απευθύνθηκαν συγκεκριμένες ερωτήσεις, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Δεν είναι και ενοφανής η συζήτηση. Τα περισσότερα στοιχεία τα είδαμε και στη μελέτη. Αυτό αποτελεί καλή βάση για περαιτέρω συζήτηση της προτάσεως. Θα δώσω το λόγο στον συνάδελφο. Ίσως μια απάντηση, λέει. Ευχαριστώ. Μια απάντηση στην ερώτηση που αφορά τις εθελοντικέ δραστηριότητε είτε είναι στο Erasmus Plus ή στο Σώμα Αλληλεγγύης. Η πρόταση καθιστά δυσχερέστατο, Δυσχερέστατη αυτή η διάκριση, διότι κάποια τμήματα της Ευρωπαϊκής Θελοντικής Υπηρεσίας παραμένουν στο Erasmus Plus, Κυρίω για τις χώρε εταίρου και τι χώρε ΕΖΕΣ. Άρα είναι δυσχερέστατη κατάσταση για τους ετούντες. Στη Γερμανία έχουμε πολλές αιτήσει, πολλούς οργανισμούς που εργάζονται με ΜΚΟ εντός Ευρωπαϊκής Ενώσεως και εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως, χωρίς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η διάκριση μεταξύ Εράσμους Πλώ και δραστηριοτήτων του Σώματος Αλληλεγγύης σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνουν αίτηση για διαφορετικά προγράμματα. Οπότε περιπλέκονται τα πράγματα, αυξάνεται η γραφειοκρατία και είναι δυσχερέστατο για μας να παρουσιάσουμε την όλη κατάσταση. Άρα θα ζητούσα μεγαλύτερη πρωτοβουλία όλες οι δραστηριότητες εθελοντικές να ενταχθούν σε ένα πλαίσιο. Στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης να υπάρχουν κάποιες δραστηριότητε που απομένουν στο Erasmus Plus που είναι ισχυρότατε. Οι ανταλλαγέ μεταξύ νέων, κινητικότητα προσωπικού, υποστηρικτικέ δραστηριότητε για τους νέους, αλλά χρειάζεται διάκριση μεταξύ διαφορετικών προγραμμάτων όπου κάνουν τις δραστηριότητε είναι, ασχολούνται με τις παρόμοιες δραστηριότητε, είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Ευχαριστώ κύριο Σταντίνα. Θα ήθελα να επαναλάβω αυτά που είπε ο Μάνφρεντ πρέπει να συγκεντρωθούν οι δραστηριότητες όλες εντός του Erasmus Plus. Αλλιώς διατρέχουμε τον κίνδυνο πολλαπλών προγραμμάτων χωρίς διασύνδεση μεταξύ τους. Και το άλλο, η απάντηση που αφορά το άλλο θέμα. Αν παραμένει ο κλάδος στην απασχόληση όχι. Προτιμούμε να ενταχθεί κάπου αλλού. Σε υφιστάμενα προγράμματα. Αν οι τοποθετήσεις για απασχόληση και ε, μαθητεία παραμείνουν εντό του σώματος αλληλεγγύη, η ΟΚΕ θέλει να τηρούνται τα ποιοτικά πρότυπα, η αμοιβή να ταιριάζει με την εκείνη για τα ημερομίσθια και με τις συλλογικέ συμβάσεις. Ταυτόχρονα υποστηρίζουμε υποχρεωτική σύμπραξη με μη κερδοσκοπικού οργανισμούς και φορεί, διότι αυτό μπορεί πραγματικά να εξασφαλίσει ποιότητα και να καλύψει και αυτά που είπε η Γκαμπριέλα σωστικά. Ευχαριστώ πολύ. Εσύ έχει το λόγο. Η κυρία Σίβικο. Ευχαριστώ πολύ. Σε έναν ιδανικό κόσμο δεν θα είχαμε ένα πρόγραμμα που ε, θα επικεντρώνα στην αλληλεγγύη με συμμετοχή από κερδοσκοπικές οργανώσεις. Ε, εμείς ε, θεωρούμε ότι θα πρέπει να συμμετέχουν αλλά όχι άμεσα. Σε έναν ιδανικό κόσμο όπως είπα δεν θα υπήρχε κάτι τέτοιο. Δεν θα υπήρχε ανάγκη δηλαδή κερδοσκοπικές οργανώσεις να βάζουν το χέρι τους ε, σε δράσεις αλληλεγγύης. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι αν, χρεια... αν είναι απαραίτητο να υπάρχουν και οι δύο αυτές πλευρές θα πρέπει να υπάρχει ε, σαφής διάκριση ανάμεσα στην απασχολησιμότητα και στον εθελοντισμό. Να υπάρχουν δύο σαφείς ε, τομείς, αφού δεν είμαστε σε αυτόν τον ιδανικό κόσμο που θα θέλαμε. Επίσης, θα πρέπει και οι δύο πλευρές να χρηματοδοτούνται πλήρως. Έτσι αποφεύγουμε τον κίνδυνο να υπάρχουν άνθρωποι που θα καλούν εθελοντές, ενώ στην πραγματικότητα χρειάζονται εργαζόμενους. Εμείς αυτή τη στιγμή ανησυχούμε πάρα πολύ ότι θα υπάρξουν περιπτώσεις όπου άνθρωποι θα κληθούν να παρέχουν εθελοντικές ε, υπηρεσίες ενώ στην πραγματικότητα θα καλύπτουν κανονική θέση εργασίας ή πρακτικής άσκησης. Και προσπαθούμε να λάβουμε υπόψη μας ε, στη στάση μας αυτήν την, τον, τον υβριδικό χαρακτήρα του σώματος και τη συμμετοχή των κερδοσκοπικών οργανισμών. Ε, αναφέρθηκαν κοινωνικές ε, επιχειρήσεις. Ε, θα μπορούσε να είναι μια κομψή ίσως λύση αλλά μιας και δεν υπάρχει ευρωπαϊκός ε, ορισμός για το τι ακριβώς είναι η κοινωνική επιχείρηση ούτε σε πολλά κράτη-μέλη υπάρχει τέτοιος ορισμός νομίζω ότι μια τέτοια λύση δεν είναι εφικτή. Ευχαριστώ λέει η Πρόεδρος. Επειδή ξέρω ότι ο Επίτροπος δεν έχει ε, πάρα πολύ χρόνο να μείνει μέχρι το τέλος δηλαδή σας ευχαριστούμε φυσικά για την παρουσία σας θα ήθελα να σας δώσω τώρα τον, το λόγο για να μπορέσετε και να αποχωρήσετε. I will be... Πολύ σύντομα θα σας τα πω, γιατί βρισκόμαστε στην, ε, φάση, στην πρώτη φάση των διαπραγματεύσεων. Νομίζω ότι μπορούμε να λάβουμε υπόψη μας όλα τα ζητήματα που τέθηκαν. Ας ξεκινήσουμε από τους ορισμούς διότι όπως, ε, αναφέρει, όπως ανέφερα και εισηγητικά ε, εμείς δεν θέλαμε να επιλέξουμε εξ αρχής πολύ αυστηρούς ορισμούς γιατί κάποιες φορές έρχεται η ζωή και διαψεύδει τους πολύ αυστηρούς ορισμούς που μπορεί να έχει δώσει κανείς. Γι' αυτό και θέλαμε στη, διάρκεια της υλοποίηση και έπειτα από την ολοκλήρωση της πρώτης δοκιμαστικής φάσης της πιλωτικής λειτουργίας του προγράμματος να προχωρήσουμε σε λεπτομερέστερους ορισμούς. Διότι αυτή τη στιγμή έχουμε καλή συνεργασία με μη κυβερνητικέ οργανώσεις, με, άλλες, ε, με άλλους οργανισμούς. Επομένως μπορούμε να βασιστούμε στην δική τους εμπειρία και ταυτόχρονα μπορούμε βεβαίως να βασιστούμε και στις δικές μας ε, εμπειρίες που αποκομίσαμε από την Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία. Έτσι λοιπόν καταφέραμε να καταλήξουμε σε έναν κοινό ορισμό γενικό όσον αφορά τις δράσεις αλληλεγγύης. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση, 186 ε, μάλλον ε, εκατομμύρια ευρώ. ευρώ ε, φρέσκια χρηματοδότηση. Φρέσκια όχι ακριβώς, διότι δεν βγήκε μόλις από το νομιμασματοκοπείο αυτό το χρήμα, αλλά είναι χρήματα τα οποία δεν είχαν διατεθεί και μπορούμε πλέον να τα διαθέσουμε και να τα αξιοποιήσουμε εμείς. Άρα μιλάμε για 86,2 εκατομμύρια ευρώ. Νέα χρήματα. Όσον αφορά την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, νομίζω ότι είναι σαφές ότι υπάρχει. Στην Όρτσα, για παράδειγμα, ε, όπου ήταν μία από τις πρώτες περιοχές δραστηριοποίησης του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Εκεί λοιπόν είδα ότι δημιουργείται μία, ας την πω, διεθνή κοινότητα. Αυτή ακριβώς είναι μια κοινότητα ανθρώπων από, από πολλές χώρες δηλαδή. Αυτή ακριβώς είναι η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Όσον αφορά τις κερδοσκοπικές και μη κερδοσκοπικές ε, επιχειρήσεις και οργανισμούς. Εγώ νομίζω ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα καλό συμβασμό. Αν τονίσουμε όχι τόσο τον, την νομική φύση ε, των, ε, των οργανισμών αυτών, αλλά το, την κοινωνική διάσταση των δραστηριοτήτων αυτών των οργανισμών, ακόμη και ένας κερδοσκοπικός οργανισμός μπορεί κάποιες φορές να έχει ε, πολύ σημαντικό κοινωνικό έργο και κάτι αντίστοιχο έχουμε ήδη αξιοποιήσει και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας. Είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να βρούμε μια καλή λύση με τον τρόπο που σας περιέγραψα. Όσον αφορά το, τη διάσταση της ε, απασχόλησης, ε, και το 80-70-30 που αναφέρθηκε ως αναλογία για τις δράσεις αλληλεγγύης και τις δράσεις απόκτησης επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Αυτή τη στιγμή το 100% των προσφορών αφορά την, ε, τον εθελοντισμό. Άρα πρέπει να αναπτύξουμε και να διευρύνουμε την διάσταση της απόκτησης επαγγελματικών δεξιοτήτων. Υπάρχει λοιπόν πολύ μεγάλο περιθώριο βελτίωσης σε αυτή την πλευρά του Ευρωπαϊκού Σώματος Ελληνικής. Αυτή τη στιγμή το 20% που έχουμε προβλέψει δεν είναι υπερβολικά αυστηρό, το 80% ωστόσο Νομίζω ότι είναι, είναι, είναι, από την άλλη μεριά αρκετά περιοριστικό όσον αφορά τις δράσεις αλληλεγγύης. Παρ' όλα αυτά, εμείς ε, σε κάθε περίπτωση θα προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε όσο γίνεται και όσο περνάει από το χέρι μας αυτές τις προσφορές ε, που ενισχύουν την επαγγελματική διάσταση, δηλαδή τη διάσταση της απόκτησης επαγγελματικών δεξιοτήτων. Ε, αυτά από την πλευρά μου και σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ σε όλους τους ομιλητές του πρώτου πάνελ, τον Επίτροπο Ναύρα, και περνάμε στο δεύτερο τμήμα της ακρόασης και θα παραδώσω τα ενία ε, του συντονισμού της συζήτησης στην συνάδελφο Μαριέτα Ουλφσκοκ για αυτό το δεύτερο τμήμα της ακρόασης. Well, we have... Ευχαριστώ. Έχουμε τόσα πολλά να κουβεντιάσουμε και έχουμε μείνει κάπως πίσω. Θα προσπαθήσουμε να στριμώξουμε κάποια σημεία της ημερήσιας διάταξης, ούτω ώστε όλοι να μπορέσουν να εκφραστούν. Πώς βλέπουμε εμείς τα πράγματα όσον αφορά τα θέματα αγοράς εργασίας και της απασχόλησης που μας απασχολούν στο Κοινοβούλιο. Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι σημαντικότατο να ασχοληθούμε επίσης με ασαφή ζητήματα. Αμοιβόμενη εργασία, εθελοντική και μη αμοιβόμενη εργασία ή με χαμηλή αμοιβή. Όλα είναι ένα κράμα. Και οι νέοι θα πρέπει να έχουν μια αξιοπρεπή θέση εργασίας που θα είναι αμοιβόμενη. Υπάρχουν και εκείνοι που προσπαθούν να τα προστατεύσουν αυτά τα θέματα όσον αφορά την απασχολησιμότητα των νέων. Τα χρήματα για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο που είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής Απασχόλησης και νομίζουμε ότι δεν θα πρέπει να μειωθούν οι φιλοδοξίες όσον αφορά την αξιοπρεπή απασχόληση των νέων. Θα πρέπει να ξεκινήσουν την ε, ζωή τους στον τόπο της εργασίας ε, χωρίς να αισθάνονται ότι δεν υπάρχουν σαφείς κανόνες. συμφωνούμε οι δύο επιτροπές από αυτού, αλλά είναι πολύ περίπλοκο να βρεθούν οι λύσεις τούτων λεχθέντων. Να δώσω το λόγο, εφόσον χάσαμε κάποιο χρόνο, καθυστερήσαμε, να δώσω το λόγο στους εμπειρογνώμονες που δεν έχουμε ακούσει ακόμα. Ο κ. Πιότρ Σαντόφσκι, Γενικός Γραμματέας του uh, Europe της Ευρώπης για τον Θεοντισμό να πει την άποψή του για αυτά που συζητήσαμε μέχρι τώρα και τα σχέδια για το μέλλον. Ευχαριστώ. Για να είμαι ειλικρινής, στο δεύτερο πάνελ δύσκολο να πει κανείς καινούρια πράγματα. Πολλά από αυτά που συμπεριλαμβάνω στην παρουσίασή μου έχουν αναφερθεί. Εντάχει να πω το εξής και μετά θα αναφερθώ και στην πρόσβαση των Βρετανικών φορέων μετά το Brexit. Βλέπω τη συμπεριφορά της Βρετανικής κυβερνήσεως, αμφιβάλλω κατά πόσο η διαπραγμάτευση για τη συνεχιζόμενη πρόσβαση ε, στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και σε άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα θα αποτελέσει προτεραιότητα. Αν θέλουμε να το εξετάσουμε αυτό και θέλουμε να έχουμε ενωμένη, πρέπει να έχουμε πολύ ενωμένη φωνή της κοινωνίας των πολιτών η Volant Europe ε, έχει έδρα στη Βρετανία και το Brexit ήταν μεγάλη απώλεια για όλους μας. Για το σήμα ποιότητα, το σήμα. Εξέτασε Σάιμον κατά πόσο έχουμε δύο σήματα, ένα για τον εθελοντισμό και ένα για την απασχόληση και για τους δύο κλάδους και να υπάρχουν διαφορετικοί φορείς να συμμετέχουν στο εθελοντικό κλάδο, η κοινωνία των πολιτών, εθελοντικός κλάδος που όχι μόνο θα σχεδιάζει αλλά και θα παρακολουθεί τις ε, δραστηριότητες και θα ελέγχει την ποιότητα και στον κλάδο απασχόληση θα υπάρχουν και άλλοι εταίροι, συνδικάτα, ε, δημόσιες υπηρεσίες ε, ε, απασχόλησης και θα εξασφαλίζεται εκεί ότι υπάρχει σωστή εργασία, ποιοτική και όχι διάφορες θέσεις επισφαλής με κακές αμοιβέ. Τώρα να απευθυνθούμε και στους νέους, να δημιουργήσουμε δυνατότητες. Χωρίς περαιτέρω επενδύσει στο σχεδιασμό και τη συμπαραγωγή ε, στο σώμα αλληλεγγύης ε, δεν θα μπορέσουμε να φτάσουμε στους ε, νέους που είναι σε δυσχερή θέση. Και έχουμε πρόβλημα να βασιζόμαστε μόνο στην διαδικτυακή ενημέρωση και εκπαίδευση των θελοντών. Υπάρχουν και, υπάρχει και το υπόβαθρο των διαφόρων θελοντών. Λοιπόν, εθελοντισμός έναντι απασχόλησης κάποιες ποιοτικέ θέσεις ίσως αντικατασταθούν από μία αμοιβόμενη θελοντική εργασία. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Γι' αυτό θα πρέπει ε, η πρόσβαση στον κλάδο των εθελοντικών περιορίζεται μόνο στον εθελοντικό τομέα, οργανώσεις νεολαίας, ε, κοινωνία των πολιτών, αλλά και στον ιδιωτικό τομέα. Θα λέγαμε ότι ο ιδιωτικό τομέα δεν μπορεί να συμμετάσχει στι υπηρεσίε απασχόληση. Πρέπει να υπάρχουν και άλλοι. Ε, που θα, ο ιδιωτικό τομέα συμμετέχει, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν και τα συνδικάτα ε, και άλλοι που θα ελέγχουν την ποιότητα των θέσεων απασχόληση που προσφέρονται και τι αμοιβέ. Αναφέρθηκαν οι τοποθετήσει ε, και όσον αφορά την πρόληψη των καταστροφών. Το πρόγραμμα τη Ευρωπαϊκή Ενώση για του Εθελοντέ δίνει έξοχε δυνατότητε για του νέου και σε όλου του εθελοντέ όλων των ηλικιών πάνω των, από 18 και πάνω από 30 για την πρόληψη των καταστροφών εκτός των σύνορων τη Ευρωπαϊκή Ένωση να συμμετάσχουν. Υπάρχουν μαθήματα και πρακτικές που μπορούμε να πάρουν τους εθελοντές και να ληφθούν υπόψη στο Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντισμού. Δυστυχώ έφυγε ο κ. Βουλευτή που είπε αυτό που θέλω να αναφέρω. Δεν θα έβαζα το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύη, του τους εθελοντέ να ανταποκρίνονται άμεσα σε μια καταστροφή. Εδώ χρειάζονται πολύ καλά εκπαιδευμένοι εθελοντέ και προσωπικό. Ε, αυτοί πρέπει να χρησιμοποιούνται. Και όχι οι νέοι που ίσω να έχουν και μειονεκτικό υπόβαθρο και θα πρέπει να διατρέξουν ε, κινδύνους. Έξι μήνες μετά την καταστροφή, εντάξει, μπορούν να πάνε να βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση, ε, και να τονώσουν το ηθικό των κοινωνιών. Θα φτάσουμε σε 100.000 συμμετέχοντες το 2020. Αν δεν έχουμε διάφορους εμπλεκόμενους φορείς, αυτό θα είναι δύσκολο. Σε αυτό το πλαίσιο ε, θα θέλαμε να ζητήσουμε το όριο ηλικίας να πάει στα 16. Διότι έτσι όχι μόνο θα έχουμε συμμετοχή περισσότερων νέων, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν γίνεται κανείς 18 και αρχίζει να είναι εθελοντής, διότι ο εθελοντισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, περιλαμβάνει άτομα που είναι κάτω από 18. Αναφέρθηκα στο ποιοτικό σήμα, μετά στα θετικά αποτελέσματα όσον αφορά την αγορά εργασίας. Ε, θα πρέπει ε, όταν εφαρμοστεί το πρόγραμμα έχουμε στόχο και τους εργοδότες ενθαρρύνοντας να αναγνωρίσουν την εμπειρία που αποκτούν οι συμμετέχοντες στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης στον εθελοντικό κλάδο, να αναγνωρίζονται οι δεξιότητες και οι γνώσεις που έχουν αποκομίσει από τον εθελοντισμό σαν πραγματικές δεξιότητες ε, που τους κάνουν αυτούς τους νέους άμεσα απασχολήσιμους. Αυτά και ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος τώρα στον κύριο Κώστα Μοσχοχωρίτη, Γενικό Γραμματέα. Συγγνώμη, είναι λίγο δύσκολο το, το όνομά σα για να το προφέρω. Έχετε το λόγο. Συγγνώμη, εγώ φταίω για το επίθετό μου, αλλά εδώ είμαι για να σα βοηθήσω. Καλησπέρα σε όλου και ευχαριστώ ε, όλους σας για την πρόσκληση που απευθύνατε στην InterSource προκειμένου να τοποθετηθούμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για ένα τόσο συμβαλικό θέμα όπως η πρωτοβουλία για το, η σύσταση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.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 Έχουμε ένα πολύ ουσιαστικό και θεμελιώδη πόρο, τους νέους, καθώς και μια βασική αρχή αξία, την αλληλεγγύη. Αυτό σημαίνει ότι η κοινωνία βασίζεται στην αμοιβαίο σεβασμό, η συνεργασία και τις κοινέ ευθύνε. Είναι σπουδαία πρωτοβουλία, ιδιαίτερα σε αυτούς τους καιρούς, όταν η αλληλεγγύη δοκιμάζεται καθημερινά και η κοινή γνώμη τίνει να στρέφεται κατά των εκφράσεων αλληλεγγύης, όπως για παράδειγμα της έρευνας και διάσωσης στην Μεσόγειο θάλασσα κάποια στιγμή όπου η αλληλεγγύη λείπει και όπου οι χώρες ακόμα κλείνουν τα σύνορά τους στους ετούντες άσυλο. Είμαι άνθρωπος και νομίζω πως τίποτα από ότι είναι ανθρώπινο, δεν, είναι, δεν μου είναι ανίκιο ή ξένο. Ε, νομίζω πως αυτή είναι μια αρχή που τονίζει την αρχή της αλληλεγγύης και καθιστά σε αυτή την στήριξή μας σε αυτή την πρωτοβουλία. Ωστόσο, ενώ αυτή η πρωτοβουλία είναι αξιέπαινη, ε, περιλαμβάνει κάποια στοιχεία που χρειάζεται περισσότερη συζήτηση και διευκρινήση. Τα περισσότερα βέβαια ήδη αναφέρθηκαν, γι' αυτό και δεν θα μακρηγορήσω. Πρώτα απ' όλα, κάποιοι ορισμοί δεν, είναι ξεκάθαροι. Ο ορισμός της ε, δραστηριότητας αλληλεγγύης και της τοποθέτησης αλληλεγγύης ε, είναι ασαφής, χρειάζονται διευκρίνηση. Ούτε επίσης ε, η σήμαση ποιότητας δεν ορίζεται ξεκάθαρα. Την άλλη πλευρά, η συμμετοχή φορέων που είναι κερδοσκοπικοί είναι ζήτημα γιατί υπάρχει ένταση ανάμεσα στην αλληλεγγύη και τη δραστηριότητα την κερδοσκοπική διότι η αλληλεγγύη τελικά μπορεί να είναι μια παροχή υπηρεσίας ε, με σκοπό το κέρδος. Ε, βεβαίως εδώ δεν αναφέρομαι στις δραστηριότητες ε, του, της ε, της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Ναι, το να συνδυάζουμε αμοιβόμενες θέσεις με τις ε, εθελοντικές θέσεις φαίνεται, μπορεί να οδηγήσει σε απομάκρυση από την αρχική πρόθεση. Οι νέοι καλούνται να εκφράσουν αλληλεγγύη τους και να βοηθήσουν αυτούς που έχουν ανάγκη ενώ ε, αποκτούν εμπειρία και δεξιότητες. Ενώ όταν κανείς πληρώνεται για μια τέτοια δραστηριότητα δεν θα είναι λάθος φυσικά αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν θα πρέπει να είναι κομμάτι της πρωτοβουλίας η πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης δεν μπορεί να είναι απάντηση βεβαίως για την ανεργία των νέων. Υπάρχουν άλλα μέσα για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Κάτι άλλο που θα πρέπει να αποσαφινιστεί αφορά τις ε, δημοσιονομικές διαδικασίες και φυσικά την ανάγκη για φρέσκο χρήμα, πράγμα που ήδη υπόθηκε αρκετές φορές. Αυτές είναι λοιπόν οι παρατηρήσεις που εγώ ήθελα να τονίσω και να πω ξανά ότι αυτή η πρωτοβουλία είναι εξαιρετική και ευχαριστώ και πάλι που μας καλέσατε να εκφράσουμε τη γνώμη μας για αυτήν την πρωτοβουλία. Thank you. Then I'll give ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στην Άννα Βίντεγκρεν που είναι Γενική Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεότητας. Mm. Σας ευχαριστώ και σας ευχαριστώ που, είσαστε, που με καλέσατε σήμερα εδώ να σας, σας δώσω τη γνώμη του φόρου μας εν γέννη καλωσορίζουμε αυτή την πρωτοβουλία γιατί στόχο έχει να δημιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες ώστε οι νέοι να μπορέσουν να συμμετέχουν σε ποιοτικές εθελοντικές εργασίες και επαγγελματικέ εμπειρίες. Είμαστε υπέρ της υπεράσπισης των ευρωπαϊκών αξιών, το ρόλο του εθελοντισμού στην ενίσχυση της κοινωνίας μας και στην ενίσχυση της επαγγελματική κατάρτισης των νέων μας. Αυτή είναι μία από τις βασικές, ε, τα βασικά πλεονεκτήματα αυτής της προτάσεις, ιδιαίτερα αφορά ε, την τοποθέτηση εντός της χώρας ή και, τη... εκτός των συνόρων. Είναι ένας δρόμος ώστε οι νέοι να μπορέσουν να συμμετέχουν σε προγράμματα που να είναι όμως ευέλικτα και προσαρμόσιμα στους νέους και τις ανάγκες τους. Ε, θα πρέπει να μπορέσουμε να αντλήσουμε εμπειρία από τις υπάρχουσες ε, οργανώσεις για να μπορέσουμε να έχουμε ποιοτικές ε, θέσεις εθελοντικές για τους νέους προγράμματα που προσαρμόζονται στις χιλιάδες εθελοντών και οργανώσεων που εργάζονται επί, τόπου καθημερινά και όχι να επιβάλλουμε εθελοντική εργασία. Οι νέοι και οι οργανώσεις των νέων θα πρέπει να είναι στην καρδιά αυτής της διαχείρισης ε, σε εθνικό επίπεδο. Επίσης, η συμμετοχή των νέων θα πρέπει να διευκολύνεται και να μπορούν δηλαδή να, να μπορούν να υποβάλουν τα προγράμματά τους άμεσα στην ε, η εκτελεστική αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η συμμετοχή των νέων θα είναι θετική, όμως υπό την πρόταση αυτή δεν υπάρχει μεγάλη συνοχή και χρειάζεται να γίνουν μεγάλες αλλαγές ώστε να μπορέσει να επιτύχει τους στόχους της. Ε, γιατί επικρατεί σύγχυση ανάμεσα σε δύο διαφορετικές πραγματικότητες και αυτό οδηγεί στον κίνδυνο να αντικατασταθούν οι ποιοτικέ θέσεις απασχόλησης από εθελοντικές θέσεις. Θα πρέπει δηλαδή η εθελοντική προσφορά να γίνεται σε, προς μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που έχουν λάβει τη σήμα ποιότητας του, του σώματος. Έτσι οι νέοι θα μπορέσουν να ωφεληθούν από αυτή την πτυχή ε, του εθελοντισμού. Τα μέτρα ποιότητας ε, θα πρέπει να ενισχυθούν, ιδιαίτερα όσον αφορά τη δημιουργία των θέσεων και να δημιουργηθούν συγκεκριμένες διαδικασίες για την απόδοση του σήματος ποιότητας. Επίση, θα πρέπει να περιλαμβάνεται σαφής ορισμός για το τι σημαίνει ποιοτική προσφορά σύμφωνα με το Σώμα για το δικαιώματο του εθελοντή, ένα μήνυμα με εισόδημα, κοινωνική προστασία και προστασία της σωματικής και ψυχικής υγείας. Πιστεύουμε ότι η πρόσβαση σε ποιοτικέ θέσει απασχόληση ή οι δυνατότητε απασχόληση είναι δικαιώματα και όχι προνόμια στο Φόρουμ Νεότητα. Και γι' αυτό και καλωσορίζουμε την πρόσκληση για νέου από, από μειονεκτικά περιβάλλοντα θα πρέπει να, όντως να υπάρχει μεγαλύτερη πρόσβαση για αυτούς τους ανθρώπους. Θα πρέπει να βασιστούμε στην ε, εμπειρία του EDS για να δημιουργήσουμε δυνατότητα πρόσβασης για ανθρώπους από μειονεκτούντα περιβάλλοντα ή για ανθρώπους με ειδικές ανάγκες. Η εμπειρία μας ειδικέ ότι η στήριξη από τους οργανισμούς πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος της εμπειρίας είναι πολύ σημαντική. Η στήριξη επίσης offline και online θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμη ώστε να μπορούν να προετοιμαστούν οι νέοι πριν και μετά την ε, ε, εθελοντική τους εργασία. Καλωσορίζουμε επίση την ανακοίνωση για νέε επενδύσει στους νέου και τι αυξημένε δυνατότητε πρόσβαση για τι οργανώσει νέων σε αυτή τη χρηματοδότηση καθώ και το, 85%, 87% ε, θα πηγαίνει στον εθελοντισμό. Ωστόσο αυτό θα πρέπει να γίνει ει βάρο προγραμμάτων που ήδη τώρα προσφέρουν πολύτιμε ευκαιρίε στους νέου, ιδιαίτερα το πρόγραμμα Erasmus+. Επιπλέον χρηματοδότηση χρειάζεται για να χρηματοδοτηθεί το υπόλοιπο του Εράσμους ε, που είναι, ε, αρχικά είχε αποφασιστεί για μη επίσημες δραστηριότητες. Οι επιπλέον πόροι είναι απαραίτητοι για να συνεχιστεί η στήριξη ποιοτικών προγραμμάτων που κάνουν οι οργανώσεις των νέων. Τέλος θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι το σώμα αλληλεγγύης θα είναι κομμάτι μιας ευρύτερης, πιο συνεχτικής και διαρκούς προσπάθειας της Ένωσης για επένδυση στη νεότητα. Δεν πρέπει να το δούμε χωριστά από άλλα προγράμματα για τους νέους, αλλά ως ένα εργαλείο για να επιτευχθεί επιτυχής εφαρμογή του επόμενου πλαισίου ε, της ε, στρατηγικής δηλαδή της Ένωσης για τους νέους, ώστε να εφαρμοστούν δηλαδή συγκεκριμένα προγράμματα δράσης για τους νέους. Είναι μια ευκαιρία για πιο συντονισμένη προσέγγιση στον εθελοντισμό στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εστιάσει στην ανάπτυξη, στήριξη και συντήρηση διυπηρεσιακής και διαθεσμικής συνεργασίας για την εθελοντισμό στην Ευρώπη, να λάβει υπόψη τους εθελοντισμού, τα δικαιώματα των εθελοντών, αλλά και των εθελοντικών οργανώσεων. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ. Άρα μπορούμε να ακούσουμε όσους θέλουν να προσθέσουν κάτι σύντομα, να υποβάλουν ερωτήσεις, να εκφράσουν σχόλια. Ο κ. Μπενιφάη, η κυρία Τρίπελ. Ο κ. Μπενιφάη. Η κυρία Τρίπελ και οι υπόλοιποι. Yes, well, it seems to me clear that είναι σαφές για μένα από τη συζήτηση ότι ακούστηκαν διάφορα επικριτικά σχόλια. Και πολλοί όμως έδειξαν ότι κατανοούν τις δυνατότητες που υπάρχει αυτό το πρόγραμμα. Για να είμαστε ειλικρινεί, είναι ξεκάθαρο, κατά την άποψή μου, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να δώσει ένα πολιτικό βάρος στην πρόταση. Νομίζω ότι θα πρέπει να κινηθούμε με ταχύτητα αλλά και με την απαραίτητη επαφή και συνομιλία με τους εμπλεκόμενους φορείς διότι είναι περίπλοκο το ζήτημα. Πρώτα απ' όλα το θέμα των πόρων. Είναι σημαντικό θέμα. Παραμένει στη συζήτηση. Άλλο θέμα πώς να συμβιβαστούμε όσον αφορά τον κλάδο της απασχόλησης. Ελπίζουμε να υπάρξει ε, κάποια συνένεση. Από ό,τι άκουσα μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο νομικό πλαίσιο. Κάτι που δεν είναι εύκολο να συνταχθεί, να γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ εκείνων που μπορεί να έχουν πρόσβαση σε διάφορες δυνατότητες. Εθελοντική δραστηριότητα και τις ευκαιρίες απασχόλησης. Το θέμα της χρηματοδότησης θα επηρεάσει κάποιες προτάσεις όσον αφορά το διαχωρισμό των πόρων για τις δύο κλάδους, απασχόληση και θελοντισμού, ε, πρέπει να τονίσουμε την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Αυτό είναι κάτι που αμφισβητείται ακόμα. Να πω και δύο πράγματα ακόμα εν συντομία. Πέρα από τα προαναφερθέντα. Κάτι ακόμα που μπορούμε να επεξεργαστούμε. Η ευρωπαϊκή διάσταση των προγραμμάτων. Σε κάποιες περιπτώσεις δεν γίνονται πλήρω αντιληπτές ακόμα και όταν κουβεντιάζουμε μεταξύ μα. Ίσως υπάρχει ο κίνδυνος να αντικατασταθούν πόροι εθνική για θελοντική δραστηριότητα με κάτι που ίσως τελικά να μην έχει υπερεθνικό χαρακτήρα. Πρέπει αυτό να αποσαφινιστεί. Σημαντικό είναι να δούμε πόσο μπορούμε να διευρύνουμε το πεδίο κάλυψη όσον αφορά τις χώρες που συμμετέχουν από την αρχή, στο βαθμό του δυνατού. Ήδη ετέθη αυτό. Και κάτι άλλο. Η πραγματική προπτική, οι δυνατότητες. Να χρησιμοποιηθούν οι ευκαιρίες για να αυξηθούν οι δυνατότητες να έχουμε έναν χώρο όπου οι νέοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ευκαιρίες. Ευκαιρίες που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν έχουμε τη νέα πρωτοβουλία, ας γίνει χρήσιμη για να διασκεδάσει μια ανησυχία που έχουν οι νέοι. Τουλάχιστον όταν μιλά μαζί τους. Λένε, πού μπορώ να βρω τις πληροφορίε για όλα αυτά που μπορώ να κάνω. Και μου προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανταλλαγές, ε, ε, εθελοντική εργασία, ευκαιρίες για απασχόληση κλπ. Πρέπει να υπάρχει μια ενιαία θηρίδα, ένα σημείο στο οποίο πάνε οι νέοι για να πληροφορηθούν. Για να λειτουργήσει καλύτερα το πρόγραμμα σε συνάρτηση ε, με όλα αυτά που ήδη αναφέρθηκαν. Η κυρία Τρίπελ, ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη που έχω φωνήσει τον Τζον Γουέιν σήμερα και όλο χειροτερεύει. Λοιπόν, κυρία Ούσκοκ, είπατε κάτι ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει μια αμοιβόμενη εργασία ή με κακή αμοιβή για κανέναν, ούτε για τους νέους. Βέβαια, αυτό θέλω να το υπογραμμίσω. Οι νέοι θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα σε αξιοπρεπή αμοιβή. Και αυτό που κάνουμε τώρα εδώ με το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύη, όπω ονομαστεί, εγώ προτείνω διαφορετικό τίτλο στο φορέα αυτό, δεν θα πρέπει να πάμε κατά του πολιτικού στόχου. Πρέπει να είναι σαφέστατο ότι δεν θα υπάρχει κατάχρηση των νέων προτινόμενων μέσων. Δεν έχω πιστεί ακόμα ότι υπάρχουν αρκετά καλοί ορισμοί για να αποφευθεί η κατάχρηση και η παρεξήγηση. Θα το επεξεργαστούμε αυτό, να δούμε αν θα βρούμε τους σωστούς ορισμούς δεν ξέρω αν θα επιμείνω στην πρότασή μου ή θα την αποσύρω. Δεν είναι ίσως δυνατό να καθοριστούν ξεκάθαρα τα όρια όσον αφορά την ε, διαδικτυακή κατάρτιση. Ε, ε, δεν ξέρω αν ταιριάζει με την κοσμοπολίτικη προσέγγιση που έχουν οι νέοι σήμερα που χρησιμοποιούν όλα τα εργαλεία τα διαδικτυακά. Τώρα όταν έχουμε νέους με προβλήματα σε μειονεκτική θέση χρειάζονται μεγάλη υποστήριξη όπως τα σχολεία. Ακόμα και αν υπάρχουν iPad και τεχνικός εξοπλισμός, το θέμα σχέσεως μαθητών και διδασκάλων είναι μέσω του αναλογικού κόσμου. Χρειάζεται λοιπόν η ανθρώπινη επαφή, όχι μόνο τα ψηφιακά εργασία. Πρέπει να τα χρησιμοποιούμε, αλλά μόνο ψηφιακά ε, ε, μέσα και διαδίκτυο δεν αρκούν. Είναι το θέμα και των ανθρωπίνων σχέσεων. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα αν υπάρχει θετικός αντίκτυπος στην αγορά εργασίας, δεν είμαι σίγουρη. Ξέρω ότι κάποιοι ελπίζουν ότι θα υπάρξει θετικός αντίκτυπος στην αγορά εργασίας. Κυρίως στις νοτιοευρωπαϊκές χώρες, όπου η εναργία των νέων είναι πολύ ψηλή. Όπως βλέπω εγώ τα πράγματα όμως είναι πολύ καλύτερο να διαχωρίσουμε τον εθελοντικό κλάδο από τα προγράμματα καταπολεμήσεως της ανεργίας των νέων. Να μην τα αναμειγνύουμε. Πρέπει να προωθήσουμε τα προγράμματα για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων. Αλλά να τα αναμίξουμε με το νέο προτινόμενο πρόγραμμα δεν είναι κάτι που με πείθει. Τώρα, αν οι νέοι με προβλήματα ε, και μειονεκτήματα, αν θα πρέπει να πηγαίνουν σε περιοχές που έχουν υποστεί κάποια καταστροφή, όχι χωρίς εμπειρία, με χαμηλή αμοιβή, δεν πρέπει να πηγαίνουν σε περιοχές που έχουν υποστεί καταστροφές. Ε, όσον αφορά λοιπόν πλημμύρες και σεισμούς, προσέξτε, δεν αναφερθήκαμε σε κάτι άλλο. Αν το όριο ηλικία πρέπει να είναι 18 ή πιο πριν. Θα πρέπει να είναι ενήλικέ. αν είναι κάποιο 16 ή 17 Είναι πολλοί νέοι, κάποιοι τελειώνουν τι σπουδέ, το κάναμε στη Γερμανία, ξεκινήσαν πολύ νωρί τι σπουδέ, αποφυτούν, έχουν πτυχίο και δεν είναι ακόμα ενήλικε, δεν μπορούσαν να υπογράψουν ένα συμβόλαιο. Πρέπει να αποφύγουμε λοιπόν να μην υπάρχει ο σωστό συντονισμό ηλικία με θέσει. Να μην, το όριο ηλικία να μην πάει χαμηλά. Για το Ευρωπαϊκό ε, Youth Forum πρέπει να καθορίσουμε ε, ποιο είναι ο ποιοτικό εθελοντισμό Θέλουμε εθελοντισμό υψηλής ποιότητας. Αυτό είναι και το όνομα του προγράμματος. Δεν μιλάμε για ανεργία, μιλάμε για αλληλεγγύη. Θέλουμε να αυξηθεί η αλληλεγγύη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό αυτού πρέπει να επικεντρωθούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η κυρία Σόντροβα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ε, θα ήθελα να επανέλθω σε ένα θέμα που τέθηκε λίγο νωρίτερα. Ε, αναφέρομαι στο ζήτημα της αμοιβόμενης εργασίας, των, της πρακτικής άσκησης, της απόκτησης δεξιοτήτων και της βελτίωσης της αποσχολησιμότητας. Όλα αυτά είναι η μία πλευρά, η άλλη πλευρά είναι ε, ο εθελοντισμός. Βρισκόμαστε σε μια κοινή ακρόαση των Επιτροπών Απασχόλησης και Πολιτισμού. Είναι προφανές λοιπόν ότι ε, το πρόγραμμα αυτό καλείται να καλύψει και τις δύο πλευρές. Άρα το, το ερώτημα που πρέπει να μας απασχολήσει είναι αν θέλουμε το πρόγραμμα αυτό να ενταχθεί στο πλαίσιο του Erasmus Plus. Εγώ σέβομαι βεβαίως τον κύριο, τον ε, κύριο Τραντίνα, αλλά αν καταλήξουμε ε, καταλήξουμε στο πλαίσιο αυτού του προγράμματο να έχουμε ανθρώπου οι οποίοι στην πραγματικότητα θέλουν να αποκτήσουν επαγγελματική ε, εμπειρία, τότε τέτοιου είδου προγράμματα πρέπει να σα πω ότι δεν είναι ε, σύνηθε να εντάσσονται στο Εράσμου. Υπάρχουν άλλα εργαλεία και άλλα, άλλοι μηχανισμοί, άλλα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας Θα μπορούσαμε να πούμε ε, καλύτερα ίσως ότι πρόκειται για δράσεις αλληλεγγύης, που στόχο έχουν την βελτίωση των δυνατοτήτων πρόσληψης, της απασχολησιμότητας δηλαδή, ε, αλλά αυτό βεβαίως θα σήμαινε ότι ένα τέτοιο πρόγραμμα θα έπρεπε να λάβει και ένα ξεχωριστό αυτόνομο προϋπολογισμό. Ε, αυτόνομο από, του, από εκείνον του Erasmus Plus βεβαίως. Ευχαριστώ. Julie Ward. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους, το Χόλγερ, για, όλους, για, για το εξαιρετικό τους έργο και θέλω να ευχαριστήσω και όλους τους ομιλητές που νομίζω ότι είπαν πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Ήταν άνθρωποι εμπειρογνώμονες με την ε, πραγματική έννοια, γνωρίζουν το αντικείμενό τους και βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της υπεράσπισης, της ευημερίας και των ε, δικαιωμάτων των νέων ανθρώπων. Η αλληλεγγύη λοιπόν νομίζω ότι είναι το βασικό θέμα και ως Βρετανίδα Ευρωβουλευτής που εργάστηκε για πολλά χρόνια με νέους και παρακολουθώντας και την καταστροφή που σημαίνει το Brexit για την ε, Βρετανική νεολαία, εγώ θα ήθελα να καλέσω αυτό το πρόγραμμα να επιδείξει αλληλεγγύη και σε νέους ανθρώπους που θα βρίσκονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γνωρίζω από το έργο μου στο Κόσοβο, στη Σερβία, στη Βοσνία Ριζιγοβίνη πόσο ε, απελπισμένοι είναι οι νέοι εκεί που λόγω του γεγονότος ότι βρίσκονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και πόσο θέλουν να ε, δημιουργήσουν επαφές και σχέσεις με ε, ανθρώπους άλλους νέους από την ε, Ευρώπη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι νέοι άνθρωποι λοιπόν στην Βρετανία αλλά και ε, σε άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης χρειάζονται την αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδίως οι νέοι που δεν ήταν και επιλογή τους το Brexit, που δεν ψήφισαν το, το Brexit, νομίζω ότι θα πρέπει να τεθούν μεταξύ άλλων στο επίκεντρο της προσοχής του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Να πω επίση κάτι σε σχέση με τη συμμετοχή των συνδικάτων. Η συμμετοχή των συνδικάτων ε, δεν, σημαίνει απαραίτητα ότι δημιουργείται ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα εργασίας. Εγώ συνεργάζομαι με πάρα πολλά συνδικάτα, για παράδειγμα με, με το Συνδικάτο των Ταχυδρομικών Υπαλλήλων στην Βρετανία που επίσης πρέπει να σας πω ότι αναπτύσσει και δικές του δράσεις αλληλεγγύης. Δεν, η δραστηριότητα των συνδικάτων δεν περιορίζεται απλώς και μόνο στην, στα εργασιακά και στα επαγγελματικά θέματα. Θα ήθελα λοιπόν να σας καλέσω, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, να έρθετε σε μεγαλύτερη επαφή με συνδικάτα για να φωτίσετε και τη δική τους οπτική. Πρόεδρος, ε, Κυρία Κώστα, έχετε το λόγο. Πιστεύω ότι βασικός κόμβος είναι η απασχόληση και θελοντισμός. Ο κίνδυνος δεν είναι μόνο αυτός που ήδη αναφέρθηκε μιας δουλειάς που αντικαθίσταται από εθελοντική δραστηριότητα, αλλά θα χάσει ο εθελοντισμός τη φύση του και σημασία σαν εθελοντισμός. Δηλαδή, σαν δωρεάν ε, παροχή αλληλεγγύης και υπηρεσίας και γίνει κάτι αμοιβόμενο. Αυτή είναι μια διάκριση θεμελιώδου σημασία που πρέπει να γίνει. Βασικό στοιχείο της προτάσεως δεν είναι ε, ένα θέμα που αφορά το 20 με 80% που λέγαμε πριν ή 30-70% είναι η φύση του σώματος που αμφισβητείται. Ε, πράγματι, η Επιτροπή Απασχόλησης έχει την αρμοδιότητα επ' αυτής της Να υπενθυμίσω. Δεν είμαι διπλωματική, τα λέω στα ίσα. Η απασχόληση ασχολείται με το θέμα του κοινωνικού, της πρόνοιας, της ένταξης, απασχολησιμότητας και της ενημέρωσης. Λοιπόν, και ο κ. Μπενιφέη το έλεγε, να δούμε έχοντας υπόψη ότι πρέπει να κατάμε το πιδάλιο, μην δημιουργήσουμε γκρίζα αγορά εργασίας, να βρούμε και αξιοπρεπή μέση λύση που διατηρεί αυτή την πτυχή παρήνει να αντέξουμε εκεί την επίσημη απασχόληση σε χώρε που δεν έχουν τέτοια ρύθμιση. Να πω και κάτι άλλο. Θα ήθελα στο τέλο τη διαδικασία, όπω είπε κάποιο, να υπάρχουν δύο μεγάλοι στόχοι. Ο πρώτο είναι να μπει στο επίκεντρο ο εθελοντισμό, όπω το περίφημο έγγραφο του 2011 που ζητούσαμε τη Λευκή Βουλή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό δεν έγινε ποτέ. Στο καθεστώ του εθελοντισμού κλπ. να επεκταθεί. Απ' την άλλη, πιστεύουμε ότι ο εθελοντισμός θα πρέπει να παραμείνει μια εμπειρία που θα μπορεί να αποκτάτε και να γίνεται σε όλα τα κάτι μελη και να εφαρμόζεται ε, και στα κάτι μελη Τα μισα κάτι κράτη-μέλη δεν έχουν νομοθεσία για τον θελοντισμό. Λοιπόν, ε, ε, θα πρέπει, θα, δεν θα πρέπει να γίνεται αντικατάσταση. Αυτό πρέπει να προσέξουμε. Τα κράτη-μέλη δεν θα πρέπει να προσφέρουν στου νέου τη δυνατότητα ε, θελοντισμού σε εθνικό επίπεδο, να δίνουν τον θελικό θελοντισμό σε εθνικό επίπεδο, αλλά να υπάρξει αλληλεπικάλυψη με την ευρωπαϊκή προσέγγιση. Λοιπόν, με τα λίγου ευρωπαϊκούς πόρους, να μην βγάλουμε τα κάστανα από τη φωτιά. Δεν ξέρω πώ μεταφράζεται αυτό, να βγάζουμε τα κάστανα από τη φωτιά για τις χώρες εκείνες που δεν θέλουν να προωθήσουν στη χώρα τους τον εθελοντισμό ή το κάνουν σε ελάχιστο βαθμό με ευρωπαϊκούς πόρους. Δεν θα συμφωνούσα. Δεν κάναμε έτσι μια δράση ευρωπαϊκή, ευρωπαϊκή διάσταση και εντός της χώρας θα πρέπει να διατηρείται ξεχωριστά ως ευρωπαϊκή. Να φαίνεται ότι είναι ευρωπαϊκό σώμα αλληλεγγύης. Είναι σημαντικότατο αυτό να ξεχωρίσει. Υπάρχει διαχωρισμός με, τους, με τον εθνικό εθελοντισμό. Ε, Πέτρα Κάμερβερτ. Κάμερβερτ. Ε, ευχαριστώ πολύ. Δεν δηλώθηκα ως πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού, ως απλή ομιλήτρια ζήτησα να μπω στον κατάλογο ομιλητών. Αυτό που συνειδητοποιώ όλο ένα και περισσότερο αυτές τις ε, δύο ώρες ε, που διαρκεί αυτή η ακρόαση είναι ότι υπάρχει αυτή η μεγάλη ανησυχία ανάμεσα στη διάκριση, μάλλον, όσον αφορά τη διάκριση ανάμεσα στον εθελοντισμό και την ε, ενίσχυση ε, της ε, απόκτησης επαγγελματικών δικαιωμάτων, δεξιοτήτων. Συγγνώμη. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να μας απασχολήσει. Να μην οδηγήσει δηλαδή ο εθελοντισμός στην υποκατάσταση, στη χειρότερη περίπτωση, κανονικών θέσεων εργασίας. Λοιπόν, ίσως από, έχοντας κατά νου αυτά θα μπορούσαμε να, να δούμε τα εξή. Παίρνουμε την πρόταση της Χέλγκα Τρούπελ, αφήνουμε την αλληλεγγύη να παραμείνει αλληλεγγύη, να την αφήσουμε και να την εναποθέσουμε μάλλον ε, για, όπως το κάναμε μέχρι τώρα στην εθελοντική, ε, Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία αφενός και αφετέρου όσον αφορά την επαγγελματική ενίσχυση ε, τη βγάζουμε τελείως από το σώμα αλληλεγγύης αλλά περνάμε τα κονδύλια και τα προγράμματα αυτά στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Εγγύηση για τους Νέους που από ό,τι έχω καταλάβει είναι το κατεξοχήν εργαλείο με το οποίο θέλουμε να καταπολεμήσουμε την νεανική ανεργία ιδίως στις χώρες του Νότου της Ευρώπης. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι σοβαρή τροφή για σκέψη. Τι μπορούμε να κάνουμε για την πρακτική άσκηση, για τις μαθητείες, για την είσοδο στην, ε, στην επαγγελματική ζωή ενός νέου ανθρώπου, ε, όπου υπάρχουν ε, διάφορα συστήματα ε, αμφιλεγόμενα και υποαμοιβόμενα για πολλούς νέους ανθρώπους. Δηλαδή, λέω, να ξεχωρίσουμε δύο τομείς. Η αλληλεγγύη είναι αλληλεγγύη, αφενός αφετέρου θέλουμε να ενισχύσουμε τόσο πολύ το, την εγγύηση για την νεολαία με τέτοιο τρόπο ώστε πράγματι οι νέοι άνθρωποι να λαμβάνουν προσφορές και ευκαιρίες που θα υπερβαίνουν μάλιστα ακόμα και τις μεγαλύτερες και τις υψηλότερες δυνατότητες που θα μπορούσε να τους προσφέρει ο εθελοντισμός και κάποιο σώμα αλληλεγγύης. Νομίζω ότι αυτό που θα κριθεί στο τέλος, αυτό που θα κρίνει μάλλον την επιτυχία μας στο τέλος είναι το κατά πόσο θα μπορέσουμε να επιτύχουμε αυτήν την διάκριση ανάμεσα στον εθελοντισμό και την ε, απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων. Και βεβαίως κρίσιμο ζήτημα θα είναι και ο έλεγχος. Πώς θα ελεγχθούν όλα αυτά ε, στο τέλος στα 27 ε, κράτη-μέλη. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι ζητήματα που πρέπει και μπορούν να απασχολήσουν και τους εμπειρογνώμονες που είχαμε σήμερα εδώ μαζί μας. Ο κύριος Τραντίνα. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι αυτή θα μπορούσε να είναι μια από όλε τι λύσει και γι' αυτό λέμε στην ΟΚΕ ότι θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε τη διάσταση της αλληλεγγύης σε άλλα ήδη υπάρχοντα προγράμματα. Και εάν μιλάμε για το Erasmus Plus, υπάρχει ήδη το Erasmus Pro που ε, καλύπτει ας πούμε τις, ε, την πρακτική εξάσκηση, τις μαθητείες. Δεν υπάρχει ανάγκη δηλαδή να βγάλουμε ολόκληρο το σύστημα αυτό EDS από το Erasmus Plus και να κινδυνεύσουμε να χάσουμε ένα μεγάλο εκπαιδευτικό κομμάτι. Φυσικά η επιλογή είναι δική σας. Όταν εγώ ζητούσα, ε, ρωτούσα από τους ε, εργοδότες ε, τι νομίζουν, εκείνοι ρωτούσαν τι υπάρχει και ποιο είναι το κίνητρο για τους εργοδότες αν δεν καλύπτεται καν το κόστος. Φυσικά οι εργοδότες αναμένεται να προσθέσουν κάτι παραπάνω αλλά σίγουρα δεν ε, διευκολύνεται και η ζωή τους. Και εγώ μάλιστα εξεπλάγινο ο ίδιος που οι κοινωνικοί εταίροι μου ζητούσαν ότι να βγει ολόκληρο εκείνο το κομμάτι που αφορά την απασχόληση. Γιατί πέρα από όλες τις πρακτικές δυσκολίες, το θέμα της σύγχυσης του εθελοντισμού με την απασχόληση είναι πολύ σοβαρό. Μάλιστα. Να δώσουμε το λόγο και στον κύριο Μοσχοχωρίτη, που είναι ο Γενικός Γραμματέας της Ίντουσος. Εγώ δεν έχω πολύ περισσότερο να προσθέσω από αυτά που είπε ο προηγούμενος ομιλητής. Πρέπει νομίζω σαφώς να κάνουμε διάκριση ανάμεσα στις δύο ε, κατευθύνσεις. Για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ προέρχομαι από ανθρωπιστική οργάνωση και βλέπω την ανάγκη επικράτησης του πνεύματος αλληλεγγύης και του πνεύματος του εθελοντισμού, ενώ αντίθετα από την άλλη πλευρά τον ε, επαγγελματισμό δεν θα πρέπει να αναμειχθούν ε, σε αυτή τη φάση η απασχόληση με τον εθελοντισμό. Και συμφωνώ επίσης με τα όσα υπόθηκαν ε, ότι στις ε, οξύες φάσεις ε, μιας επίγουσας κατάστασης ποτέ δεν στέλνουμε ένα θελοντή. Ποτέ δεν στέλναμε θελοντή στη Σομαλία, ας πούμε, σήμερα. Υπάρχουν σοβαρές διακρίσεις που πρέπει να ε, υπάρχουν διαρκώς ε, στην άκρη του μυαλού μας. Ναι, μια σύντομη παρατήρηση. Ίσως θα πρέπει όντω να γίνει μια πιο ισχυρή και πιο σταθερή διάκριση ανάμεσα στον εθελοντισμό και τις θέσεις απασχόλησης γιατί θα πρέπει να υπάρξει καλύτερη ορισμός του τι είναι εθελοντισμός. Σήμερα είναι πολύ στενός ο ορισμός. Έχουμε το βασικό έγγραφο του 11 που εξακολουθεί να ισχύει και ο εθελοντισμός υπάρχει σε τυπικό και άτυπο επίπεδο. Ε, αυτό θα πρέπει να είναι σαφές στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, ώστε να δημιουργηθεί και καλύτερη διάκριση ανάμεσα στις δύο κατευθύνσεις. Το ποιοτική, ποιοτικός εθελοντισμός δεν συμβαίνει έτσι απλά ο εθελοντισμός, πρέπει σωστά να σχεδιαστεί και όλοι νομίζω πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Δεν είναι δωρεάν τελείως όλη αυτή η προσπάθεια. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ και τώρα θα δώσω και πάλι την Προεδρία Α, θα δώσω συγγνώμη. Το λόγο πάλι στην Άννα. Μάλιστα, ευχαριστώ. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει σαφήνεια γιατί αυτό διαφορετικά είναι κίνδυνος ε, για τις ποιοτικέ ε, θελοντικές θέσεις και την αντικατάσταση θέσεων, ποιοτικών θέσεων απασχόλησης από εθελοντές. Διάκριση λοιπόν μεταξύ των ε, δύο ορισμός της ποιοτική εθελοντικής θέσης, όλα αυτά είναι πολύ επιτακτικές ανάγκες και τέλος να πω ότι Θα πρέπει να έχει αρκετούς σπόρους αυτό, αυτή η προσπάθεια, αλλά ε, και στην διαχείριση και παρακολούθηση θα πρέπει να συμμετέχουν δηλαδή οργανώσεις των ε, νέων και οι οργανώσεις που εφαρμόζουν, τις, που τοποθετούν τους εθελοντές, γιατί διαφορετικά δεν θα επιτευχθούν οι στόχοι. Ευχαριστώ, κύριος Φανχέμπελ. Σας ευχαριστώ. Ίσως να μην εξαρτάται από μένα, το τι θα μπει ακριβώς στο πρόγραμμα, αλλά κάποιες σκέψεις μόνο. Πρώτον, νομίζω ότι αν ξαναδούμε την αρχική στιγμή, της δήλωσης ε, για την κατάσταση στην Ένωση και την αλληλεγγύη ήταν ακριβώς μετά το Brexit και έπρεπε να τονιστεί το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Συνοχή και η Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη βρίσκονται στην, στον πυρήνα της Ένωσης. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό και αυτή είναι η καρδιά αυτού του ε, σώματος. Το να τα αναμειγνύουμε με άλλα θέματα μπορεί να κάπως να διαχέει και να... Ε, ε απομακρύνει από αυτή την αρχική ιδέα. Και κάτι ακόμα, συζητούσαμε την αγορά εργασία ή την δυνητική επιρροή αυτού του προγράμματος στην αγορά εργασία. Μα το πρόγραμμα αυτό δεν είναι πολύ μικρό για να πούμε ότι θα έχει σημασία σε σχέση με την αγορά εργασία, Ακόμα και το Erasmus Plus. Μπορούμε να μιλήσουμε για επιρροή του Erasmus Plus στην αγορά εργασία. Είναι εξαιρετικά ισχνή για να πούμε ότι επηρεάζει την αγορά εργασία. Άρα λοιπόν ίσω και να είναι συμβολικό το να έχουμε την πτυχή της απασχόλησης στο πρόγραμμα. Επίσης είναι αρκετά σαφές ότι οι νέοι μαθαίνουν πολλά από την εθελοντική τους δραστηριότητα, ειδικά και συμφωνώ απόλυτα με την Πέτρα, όταν δηλαδή μπορούμε να έχουμε ποιοτική εθελοντική εργασία, τότε η, μάθηση είναι βαθιά και πολύ ε, ε, ποιοτική. Αυτού του είδους η εκμάθηση και η απόκτηση δεξιοτήτων έχει μία πτυχή που επηρεάζει την δυνατότητα απασχόλησης αργότερα των νέων αυτών. Το χρησιμοποιούν μετά για να μπορέσουν να βρουν θέσεις δουλειάς. Ε, Τελευταία παρατήρηση δεν ξέρουμε ακριβώς τι ακριβώς είχε κατά νου ο κύριος Γιούγκερ που κατέθεσε αυτή την πρόταση. Δική μας δουλειά όμως είναι να δούμε ε, τι είναι τελικά εφικτό. Εσείς μιλήσατε τώρα για την απασχόληση των νέων. Φυσικά είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα αυτό. Ταυτόχρονα όμως ε, θα πρέπει να μας απασχολήσει και η δημιουργία ε, ενός εργαλείου ε, που θα προσφέρει κάτι νέο, ε, κάτι που θα είναι διαφορετικό από τα υπάρχοντα εργαλεία μας. Ακόμη και αν αφορά την είσοδο των νέων στην αγορά εργασίας. Αυτά από μένα και να παραδώσω τώρα στην Πρόεδρο της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας. Ευχαριστώ πολύ. το λόγο έχει ζητήσει η Χέλγα Τρίπελ. Ευχαριστώ. Από την αρχή της συζήτησης σήμερα το απόγευμα είχα πει ότι θέλω να τονίσω ότι ε, είναι ανάγκη να καταπολεμηθεί η νεανική ανεργία, αλλά δεν θα πρέπει το θέμα αυτό να το μπερδέψουμε με το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Και Πίτερ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που το ξεκαθάρισες ότι πρέπει πραγματικά να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες σε αυτό το θέμα. Ε, πρέπει και δημοσιονομικά να, γίνουν, να αναλυθούν περισσότερες πρωτοβουλίες, ε, να γίνουν περισσότερες προσπάθειες, αλλά όχι μέσω αυτού του σώματος αλληλεγγύης. Κατανοώ ότι, πρέπει, ε, ότι θέλεις περισσότερη αλληλεγγύη λόγω και της κατάστασης που θα ακολουθήσει μετά το Brexit αφενός. Αφετέρου όμως γνωρίζουμε πολύ καλά ότι έχουμε, έχουμε σε κάποιες χώρες 30, 20, 30 και 40% νεανικής ανεργίας και θέλουμε να, ε, να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό. Δεν ερχόμαστε σε αντίθεση με τους πολιτικούς στόχους του Συμβουλίου και της Κομισιόν. Λέμε όμως ότι θέλουμε σαφήνεια ως προς τους στόχους που θα τεθούν και να μην μπερδέψουμε τις δύο διαστάσεις. Όσον αφορά την πρόταση του, του Juncker, ε, εμείς ε, καλούμαστε να ερμηνεύσουμε τώρα την πρόταση του ε, του Προέδρου της Κομισιόν. Εγώ την επόμενη εβδομάδα έχω συνάντηση μαζί του και θα το ρωτήσω ποια ακριβώς είναι η πρόθεση ε, που έχει ε, όσον αφορά την σύσταση αυτού του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Γιατί δεν νομίζω ότι δεν αρκεί να πούμε απλά ότι εντάξει ωραία ιδέα αυτή του Προέδρου, ας δούμε πώς θα την εφαρμόσουμε. Νομίζω ότι καθήκον μας είναι να ξεκαθαρίσουμε τι θέλουμε να επιτύχουμε εμείς και εδώ έχουμε όλες τις δυνατότητες να διαδραματίσουμε ένα πραγματικά χρήσιμο πολιτικό ρόλο. Ευχαριστώ πολύ. Δικό μας καθήκον είναι λοιπόν να ερμηνεύσουμε και από εκεί και πέρα βεβαίως να διαμορφώσουμε με τόση σαφήνεια την πρόταση ώστε να ξέρει ο κάθε ένας, κάθε Ευρωπαίος πολίτης τι ακριβώς τελικά θα αφορά και θα περιλαμβάνει αυτός ο, ε, αυτός ο κανονισμός. Θα ήθελα να ρωτήσω την Κομισιόν αν θέλει να προσθέσει κάτι. Ναι, ευχαριστώ πολύ που μου επιτρέπετε να κάνω κάποια σχόλια και κάποιες ε, ε Θα το κάνω αυτό βεβαίως ε, συμπληρώνοντας τα όσα είπε στις απαντήσεις του ο Επίτροπος Ναυρασίτς ε, όσον αφορά τον εθελοντισμό, την απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων κτλ. Σκοπός της πρωτοβουλίας μας πάντως είναι να καταβληθεί μια μεγαλύτερη προσπάθεια γύρω από, τον, από την ελληνική στην Ευρώπη και ταυτόχρονα να ενισχύσουμε το θεματολόγιο για, την, για τους νέους στην Ευρώπη. Έπειτα από ψήφισμα λοιπόν του Ευρωπαϊκού ε, Κοινοβουλίου που είχε ζητήσει να υπάρχει μια ενιαία θηρίδα για τις δράσεις αλληλεγγύης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πνεύμα αυτό λοιπόν εντάσσεται η πρότασή μας αυτή. Προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε μια ισχυρή πρωτοβουλία η οποία θέλουμε να δίνει ευρύτερες και περισσότερες δυνατότητες στους νέους ανθρώπους. Και γι' αυτό και ε, ε, προτείνουμε αυτή την επαγγελματική διάσταση αλλά και ε, νέες μορφές εθελοντικής δράσης. Να ε, ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα. Ακούστηκαν, κάποια, ακούστηκαν διάφορα ερωτήματα ιδίως όσον αφορά το σήμα ποιότητας και τα λοιπά. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι μιλάμε ήδη για την φάση υλοποίησης υπάρχουν ορισμένα θέματα που μόνο τότε μπορούν να ξεκαθαριστούν. Φυσικά χρειάζεται ο κανονισμός να θέτει ένα σωστό πλαίσιο, αλλά η φάση της υλοποίησης θα μας δώσει τη δυνατότητα να μιλήσουμε με όλους τους φορείς, τους φορείς υλοποίησης και τους εμπλεκόμενους φορείς, ε, πώς θα ε, ε, ε, εφαρμόσουμε στην πράξη διάφορα θέματα. Βεβαίω, εκ των προτέρων μπορούμε να δημιουργήσουμε το πόρταλ, να ξεκαθαρίσουμε το τι θα περιλαμβάνουν οι κύκλοι εκπαίδευση και κατάρτιση, ποιε ακριβώ μέθοδοι εξασφάλιση, διασφάλιση τη ποιότητα θα εφαρμοστούν. Όλα αυτά βεβαίω ε, είναι σημαντικά, δεν χρειάζεται όμω να, περιγράφονται με κάθε λεπτομέρεια στον κανονισμό. Όπω υπόθηκε, βασιζόμαστε στην 20η εμπειρία τη εθελοντική υπηρεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίως έχουμε εξαίρετου εταίρου στου εθνικούς φορείς. Καθημερινή είναι η επαφή μα με του εθνικού φορεί και τι εθνικέ υπηρεσίε. Και σα το λέω ξεκάθαρα. Σα εμπιστευόμαστε, έχουμε εμπιστοσύνη, γιατί γνωρίζουμε ότι έχετε αποδείξει στην πράξη εδώ και 20 χρόνια ότι ξέρετε να αντιμετωπίζετε τι προκλήσει και τα προβλήματα που, που ανακύπτουν. Όσον αφορά την υποστήριξη. Νομίζω ότι πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το θέμα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια παρεξήγηση, αλλά όσον αφορά την φιλοξενία και την, και την ε, υποστήριξη της ε, οργανώσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτό τον, τον, τομέα. Εγώ δεν θέλω να εμείς δεν θέλουμε να εξαιρέσουμε αυτού του είδους οργανώσεις. Αντιθέτως θέλουμε να βελτιώσουμε τη συμβολή αυτών των οργανώσεων, των υποστηρικτικών. Και φυσικά η υποστήριξη αυτή δεν μπορεί να, να αφορά μόνο τα διαδικτυακά εργαλεία. Πρέπει να υπάρχει και καταπρόσωπο εκπαίδευση, ακόμη και, και ε, αποστολή ε, εκπαιδευτών σε χώρες. Όσον αφορά την ε, υλοποίηση προγραμμάτων εντός μιας χώρας και την ευρωπαϊκή διάσταση. Φυσικά, εγώ συμφωνώ. Δεν χρειάζεται να υποκαταστήσουμε εθνικά προγράμματα. Τα ευρωπαϊκά κονδύλια μπορούν να διατεθούν μόνο όταν υπάρχει πραγματικά λόγος και ανάγκη να ενισχυθεί ε, μια δραστηριότητα. Σε κάθε περίπτωση φυσικά, όπως είπατε και εσείς, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ευρωπαϊκή διάσταση αυτού του σώματος, των δραστηριοτήτων αυτού του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Φυσικά, λέει η Πρόεδρο, αλλά ξέρετε ότι όταν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ακούμε τον όρο εκτελεστική πράξη, εκτελεστικό κανονισμό, ε, φοβόμαστε πάντοτε, ε, επαγρυπνούμε, γιατί φοβόμαστε ότι η Κομισιόν θα πάρει διάφορε πρωτοβουλίε χωρί να διαβολευτεί μαζί μα και χωρί να γνωρίζουμε τι σκοπού έχει. Γι' αυτό και θέλουμε τα πράγματα να ξεκαθαριστούν σε, με τόσε πολλέ λεπτομέρειε ακόμη και αν αυτό πονάει λίγο την Κομισιόν, να μην τις αφήσουμε, αυτός είναι ο τελικός μας στόχος, να μην τις αφήσουμε πολλές, πολλά περιθώρια ερμηνείας ε, ή ελιγμών. Αυτή είναι πάντοτε η στάση του Κοινοβουλίου ε, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι θα μπορούμε πάντοτε με βάση τις δικές μας αποφάσεις να παρεμβαίνουμε και να μην μας θέτεται ε, ενώπιον τετελεσμένων στην ε, ε, υλοποίηση διαφόρων προγραμμάτων. Γιατί κάτι τέτοιο ε, το ζήσαμε με το Erasmus Plus. Πολλά πράγματα τελικά ήρθαν σε πλήρη αντίθεση με τα όσα επιθυμούσαμε εμείς, όσα επιθυμούσε και το Συμβούλιο, αλλά παρόλα αυτά συνέβησαν. Γι' αυτό και βλέπετε, βλέπετε ότι αγχωνόμαστε όποτε έχουμε να κάνουμε μια τέτοια δουλειά μαζί σας, λίγο, και είμαστε πολύ προσεκτικοί. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι η σημερινή ακρόαση ήταν εξαιρετικά ενημερωτική, εξαιρετικά χρήσιμη για όλους μας. Ευχαριστώ όλους τους εμπεριογνώμονες που μας έδωσαν πολλές χρήσιμες πληροφορίες, σημαντικές πληροφορίες, τις οποίες και θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε στο περαιτέρω έργο μας και που νομίζω ότι μας παρακίνησαν να σκεφτούμε και από μια διαφορετική σκοπιά διάφορα ζητήματα. Αυτά ε, από μένα. Ε, βλέπω, ε, θα ήθελα τώρα να δώσω την ε, δυνατότητα στους συναδέλφους της Επιτροπής Απασχόλησης να αποχωρήσουν βεβαίως. Η Επιτροπή Πολιτισμού θα συνεχίσει το έργο της, αλλά βεβαίως αν θέλετε μπορείτε να παρακολουθήσετε τις εργασίες μας αν όχι, ε, μπορείτε να αποχωρήσετε όπω είπα. Ευχαριστώ και πάλι τους εμπειρογνώμονέ μα. Θα είμαστε σε επαφές, ιδίω αν έχετε έξυπνε ιδέε ε, τις οποίες μπορούν να βοηθήσουν και εμάς στο έργο μας. Είναι πάντοτε ευπρόσδεκτες. Χέλγα Τρούπελ είναι η συγγήτριά μας, αλλά και την Επιτροπή Απασχόλησης και την Επιτροπή Πολιτισμού πάντοτε τη βοηθούν ε, οι συνεισφορές από τους εμπειρογνώμονες. Σας ευχαριστώ και πάλι για την παρουσία σας σήμερα εδώ.